Chers collègues, bonjour. Je vous propose sans tarder de commencer. Καλημέρα Προτείνω άνευ να ξεκινήσουμε τη παρακαλώ να με συγχωρήσετε που απεσίαζα χτες, αλλά ξέρω ότι προσωπή θέλει. Ένα θέμα είχε μείνει στην ημερήσια έταξη από το χτεσινό πρόγραμμα και είναι η συζήτηση για τις κοινέ διατάξεις τα ευρωπαϊκά τομέα και κατάργηση του κανονισμού 1083-2006 εκθέση του κυρίου Κόζα και διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για το Κοινωνικό Ταμείο. Προτείνω λοιπόν σχετικά με το πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτομία. Προτείνω να δώσουμε το λόγο στους ε, αρμοδίους. Και μετά θα ξεκινήσουμε τις προφορίες, θα έρθει η ώρα τους. Ο κύριος Κώσα πρώτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να συνοψίσω τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων. Στις 19 Ιουνίου είχαμε μια συνάντηση όπου συζητήθηκε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας και είχα πει ότι ο τριμερής διάλογος έχει προχωρήσει, εξήγησε σε ποιο σημείο έχει φτάσει. Συμφωνήσαμε. Ε, και προσπάθησα να ε, δω την κατάσταση. Υπάρχουν πιέσεις ώστε το ε, κοινωνικό ταμείο να έχει στο 25%. Μετά έγινε ο τριμερής διάλογος στη συνέχεια τον Ιούνιο με παρουσία και της Προέδρου και του εισηγητή για το κοινωνικό ταμείο. Είχαμε προγραμματίσει συνεδρίαση μία ώρα, αλλά δύο μισή ώρες κράτησε αυτή η αντιπαράθεση απόψεων. Καταλήξαμε μετά σε μια προκατακτική συμφωνία και εγώ υπέβαλα το κείμενο ως τροπολογία ώστε να δουν οι συνάδελφοι ποια είναι η κατάσταση. Οι συντονιστές αποφάσισαν Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού να αντικατασταθούν από τροπολογίες των πολιτικών ομάδων. Έχουν υποβληθεί 26 τροπολογίες για τις οποίες και ευχαριστώ και βέβαια έτσι καταγράφονται και οι αποκλήσεις απόψεων στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαι υπέρ της ποσοστάς του 25%. Αλλά αυτό είναι το μέγιστο που μπορούμε να περιμένουμε από το Συμβούλιο. 23,1% θα είναι το υποχρεωτικό κομμάτι και ανάλογα με τα δεδομένα απασχόληση ενδεχομένω να δοθούν προσθήκες ε, συμπληρώματα για το κοινωνικό ταμείο. Αυτή ήταν ε, η τροπολογία υπαριθμών 1. Οι τροπολογίε υπαριθμών 2 και 3 ταυτόσιμε, η πρώτη ήταν δική μου, οι ε, επόμενε δύο των σοσιαλιστών μαζί με του Πρασίνου. Σημειώνω επίση ω ποσοστό το 25%. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι η γνωμοδότηση που είχαμε υιοθετήσει πριν από ένα χρόνο εδώ δεν έκανε λόγο για συγκεκριμένο ποσοστό, αλλά για ενδεικτική μόνο ε, ποσόστοση του 25%. Άρα βλέπω κάποια αντίφαση όταν μιλάμε τώρα για ένα ε, ακριβές ποσό, σταθερό ποσό 25%. Οι τροπολογίες 4 και 5 προκύπτουν υπό το φως ε, του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου Πρόκειται για επιστηστική βοήθεια για τους πιο φτωχούς. Η τροπολογία μου σε ένα ποσό καταγράφει τα 3,5 δισεκατομμύρια. Αλλά η συζήτηση δεν αφορούσε αυτό το θέμα. Η Πρόεδρος υπέβαλε μία τροπολογία για 2,5 συν 1 δισεκατομμύρια και εμείς ετοιμάσαμε μια συμβαστική τροπολογία των υπαριθμών α. Συμβαστική που πιστεύω ότι θα, είναι, θα σας βρει σύμφωνος. Η υπαριθμών 6 είναι μια μεθοδολογική προσθήκη για τον υπολογισμό αυτού του ελάχιστου μεριδίου. Ε, μια ακόμη παρατήρηση για το 25%. Το 23,1% μπορεί να θεωρηθεί, μπορεί να αποδειχθεί παραπλανητικό, γιατί είναι λιγότερο σαν ποσοστό από το 25%. Όμως έχοντας ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο με περισσότερη ευελιξία και πιο ευέλικτους κανόνες για την προσεχή αιτία το, το 23,1% πιστεύω ότι μπορεί να είναι λύση αποδεκτή γιατί θα έχει σαν συνέπεια μερίδιο μεγαλύτερο από αυτό της προηγούμενης επταετίας των 22,1%. Περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Merci, euh, Elisabeth Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, στον τελευταίο τριμερή διάλογο, περασμένη εβδομάδα, ανέλαβε η Λιθουανική Προεδρία και σε αντίθεση με την προηγούμενη διαπραγματευτική ομάδα έδειξε πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα πνεύματος. Μιλήσαμε για το ποσοστό του 20% για την καταπολέμηση της στόχιας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, αυτό το ιερό και όσιο 20% στο έκτο για την καταπολέμηση της στόχιας δεν ενθουσιάζει περισσότερο από το 25% ε, του Ταμείου Συνοχής που μεταφέρεται στο ΕΚΤ. είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν συνήθως τα κράτη-μέλη σε σχέση με ένα συγκεκριμένο ποσοστό για ε, αυτόν τον τομέα. Η πρωτοβουλία για τους νέους ενισχύει την εγγύηση για τους νέους. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς συνδυάζονται οι δύο δράσεις. Είναι ξεκάθαρο πλέον, ενισχύεται η εγγύηση ε, για όσους είναι στην ψαλίδα 15 έως 35 έτη. Όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα πλαίσια της εγγύησης ε, γιατί αν περάσουμε από ε, τη ψαλίδα 15 25 στην 15 30 ε, σε χώρες όπως η Ισπανία θα δούμε ότι θα διπλασιαστούν τα νούμερα διότι είναι ιδιαίτερα υψηλή, υψηλό το ποσοστό της ανεργίας για όσους είναι από 25 έως 30 χρονών. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα επικεντρωθεί στις περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων ε, είναι 25% και πάνω, όμως θα χρειαστούμε περαιτέρω διευκρινήσεις. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να προσθέσουμε ότι Μπορεί να ανέβουμε και στο 30% αν τελικά ε, υπολογιστούν όλοι οι άνεργοι αυτή τη ηλικιακή ψαρίδας 15 έως 30 ορίζοντας έτσι και το κατόφλι για τις περιοχές δικαιούχους. Αυτό ε, είναι τα αποτελέσματα του πρώτου διαλόγου με την Λιθουανική Προεδρία. Πρέπει να είναι ηχηρό το μήνυμά μας ε, και κυρίως ε, να δείξουμε ότι αυτό το 25% που ανέκαθεν υπερασπιζόμασταν εμένουμε λοιπόν σε αυτό το ποσοστό παρότι με τις διαπραγματεύσεις συμφύνει στο 23,1% θα καταλήξουμε. Σέζιο Γκουτιέρες. Ε, παρακαλώ όσοι προετοιμάζουν την ψηφοφορία να αποχωρήσουν από την αίθουσα και να το κάνουν εκτός αιθούσης γιατί είναι κέρια σημασία οι διαπραγματεύσει, είναι το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Παρακαλώ ησυχία. Σέζιο Γκουτιέρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μας εξηγήσατε πώ πάνε οι διαπραγματεύσει. Όταν είχαμε την τελευταία συνάντηση στην Επιτροπή στη Σοσιαλιστική, τον, στη Σοσιαλιστική Επιτροπή είχα πει να μην δώσει, να μην κάνει παραχωρήσεις πέραν του 20, κάτω από το 25% διότι το 25% δεν είναι μόνο θέση και της Επιτροπής μας αλλά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαμε ζητήσει και είχαμε καταφέρει αυτό να είναι θέση του Κοινοβουλίου σε πολλά ψηφίσματα που εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο. Το 23,1 δεν μας ικανοποιεί, πρέπει να σας το πω αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει απάτη στα ποσοστά, απάτη από πλευράς του Συμβουλίου όταν ε, φτάσει στο τελικό ποσοστό. Είναι γεγονός ότι μας μειώνουν, το ξέρει ο εισηγητής, αλλά η απάτη είναι ότι ε, μειώνεται η αρχική βάση τα 7 δις ή 9 δις του Connecting Europe. Άρα είναι δύσκολο να απαντήσουν ε, στην στο θέμα αυτό ότι η δημοσιονομική προοπτική των επομένων 7 ετών όταν αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων, όταν αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που θα θέλουν καλύτερη κατάρτιση εν ώψη της αύξησης ε, της φτώχειας, το βασικό εργαλείο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά τα μειώνουμε και σε ποσοστό και σε συνολικό κονδύλι. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσουμε. Πιστεύω ιδίως ότι δεν πρέπει να παραδοθούμε. Συμφωνώ με τον, με τον κύριο Κώσα, με τον Άνταμ, ότι η διαπραγμάτευση στον τρίλογο είναι κάτι δύσκολο. Φαντάζομαι ότι για να υπάρξει συμφωνία κάπου πρέπει να δώσεις. Αλλά αυτό νομίζω είναι μια κόκκινη γραμμή, μια βασική θέση. Η Επιτροπή Απασχόλησης μας δεν μπορεί να ενδώσει αυτή τη στιγμή να δώσουμε τη μάχη όχι μόνο στην Περιφερειακή Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Αξίζει νομίζω γιατί δεν είναι θέμα ιδεολογίας ή πολιτικών κομμάτων. Ένα όραμα της Ευρώπης. Ένα όραμα που η πλειοψηφία όλες οι ομάδες στην Επιτροπή την έχουμε δώσει το παρελθόν και την έχουμε υποστηρίξει το παρελθόν. Λοιπόν, προτείνω να μην πάμε πιο κάτω από το 25% που είναι σωστό και ανταποκρίνεται σε μια κοινή εικόνα για το τι χρειάζεται η Ευρώπη. Κίνγκα Κούντς, Καρή Μαντελή, να δω ποια άλλη το λόγο. Και μετά η Επιτροπή. Η Κίνγκα Κούντς. Uh, θα ήθελα σύντομα να αναφέρω κάτι. Με μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με την υπηρεσία, είχαμε ελπίσει να έχουμε 4 εκατομμύρια ευρώ για το κοινωνικό ταμείο για την εξυπηρέτηση των στόχων της απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ενσωμάτωσης. Τώρα έχουμε 10 εκατομμύρια λιγότερα. Γιατί και το Connecting Europe Facility έχει βγει από τους ε, πόρους του Κοινωνικού Ταμείου και το πρόγραμμα εγγύησης νεολαίας. Άρα μπορεί να μιλάμε για ποσοστά μένα, αλλά ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε πολύ χαμηλότερα ποσά. Είναι χαμηλά λοιπόν τα ποσά. Και βλέπουμε ότι οι προεδρίες προσπαθούν να ε, μειώσουν ακόμα περισσότερο τα ποσά. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες που εκδηλώνουν. Τα ποσά και για την κοινωνική ενσωμάτωση και την διαφυγή από τη φτώχεια φαίνεται να μειώνονται και φαίνεται ότι κάποια κράτη μπορούν ε, να εξασφαλίσουν παρέκκληση αν αντίστοιχους πόρους του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης τους αξιοποιούν ε, για τους ίδιους ε, στόχους, όπως σε παραδείγμα την κατασκευή υποδομών, οδών κτλ. Ε, βλέπουμε ότι δυστυχώς υποβαθμίζονται οι φιλοδοξίες μας. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης πάντα όταν μιλούμε για την ανεργία, τα κοινωνικά προβλήματα και γι' αυτό πρέπει η Επιτροπή μας να αγωνιστεί ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό ποσό που θα καλύπτει τα εξυπηρετή του στόχους. Merci, Madame la Présidente. Ε, Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την αποσχόληση των νέων, καταρχάς μας πετάνε στο τραπέζι 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την εγγύηση νεότητα. Στην τελευταία σύνοδο κορυφής μας, κάνουνε, μας λένε ότι δεν θα είναι 6, θα είναι 8. Έρχεται η Επιτροπή και μας λέει στο ανάμεταξύ ότι τα 6 θα είναι σε μια διάρκεια 2 ετών. Όλα στα 2 χρόνια θα συγκεντρωθούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας μακροπρόθεσμος στόχος. Μετά από 2 χρόνια. Τι γίνεται αν δεν έχουμε χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, τα ποσά δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Το ότι δεν αντιδράσαμε στην ανεργία νέων τα τελευταία χρόνια δείχνουν οι έρευνε ότι μα τύχησε 50 δι. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασία λέει ότι για να υπάρξει μια νέα δυναμική χρειαζόμαστε 21 δι. Η ερώτησή μου είναι πώ θα χειριστούμε αυτά τα δύο δι που εμφανίζονται δεν ξέρω από πού και που σήμερα δεν λαμβάνονται υπόψη στην ουσία στις διαπραγματεύσεις. Αυτό, αυτή την εντύπωση έχω. Ευχαριστώ. Πρώτον, να ευχαριστήσω πολύ τους, τον εισηγητή μας, Άνταμ Κόσα, διότι καταφέραμε και κάναμε μια πολύ καρποφόρα διαπραγμάτευση Σήμερα μας έχει ζαλίσει αυτό το, ποσοστό, αυτό το θέμα των ποσοστών, θα, θα επανέλθουμε. Πριν συζητήσουμε για τα ποσοστά, είχαμε όμως μια πρώτη νίκη εναντί του Συμβουλίου, που είναι η αρχή του ότι αυτό το κομμάτι δεσμεύε, είναι, γίνεται δεσμευμένο στα πλαίσια του κοινωνικού ταμείου. Με θεματικούς στόχους, χάρη στην αποφασιστικότητα του εισηγητή, κερδίσαμε ένα ποσοστό στο κοινωνικό ταμείο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας. Δεύτερον, το κομμάτι που κερδίζουμε σε σχέση με το μεταξύ, μεταξύ του υφιστάμενου ποσοστού του κοινωνικού ταμείου και του στόχου δεν καθορίζεται από την φύση των εμπλεκόμενων περιφερειών αλλά με βάση το ποσοστό απασχόλησης που σημαίνει το κριτήριο προσαρμόζεται απόλυτα στην κοινωνική βάση του κοινωνικού ταμείου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και εκ νέου ευχαριστώ τον εισηγητή. Ωστόσο αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι στην Επιτροπή ζητούν από τη διαπραγματευτική ομάδα να είναι πιο σκληρή και να επανέλθει στην αρχή του 25%. Εγώ είμαι υπέρ και θέλω να δώσω ένα τελευταίο επιχείρημα υπέρ αυτού. Το Κοινοβούλιο ψήφισε, έδωσε καταρχήν συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρω ότι για πολλούς συναδέλφους ήταν δύσκολο. Ξέρουμε ότι ο προπολογισμό δεν είναι στο ύψος των προκλήσεων της Ένωσης υπάρχουν κάποια πολύ κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να ψηφίσουμε και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πολιτική συνοχής. Το αποθεματικό επί, ε, επίδοσης ή του, την θέση όλων μακροοικονομικών επιδόσεων. Δεν είμαι βέβαιος, βέβαιο ότι το Κοινοβούλιο θα έχει όλο το περιθώριο διαπραγματευσής που πρέπει να έχει. Εάν εμείς πετύχουμε εδώ στην Επιτροπή μια ευρεία συνένεση για περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης μέσω των πολιτικών μας στόχων θα γίνει έξω από το κοινωνικό ταμείο, ανεξάρτητα από αυτά που θα αποφασίσει η Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά για τη συζήτηση. Για την έκθεση τώρα για τον κανονισμό του κοινωνικού ταμείου αυτή καθεαυτή, οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει με την Λιθουανική Προεδρία μας δίνουν ελπίδες να κλείσουμε υπό δύο σε, σε καλές συνθήκες. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή Εμμανουέλ Γκελάνγκ, για να συμβάλλει στη συζήτηση και μετά θα σας δώσω το λόγο ξανά στον εισηγητή. Κύριε Γκελέν. Καλημέρα. Α, το ποσοστό 23,1 αντί για το 25%. Είναι μεγάλη απώλεια για την επένδυση σε ανθρώπινους φόρους που δύναται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφής η αύξηση σε σχέση με την τωρινή περίοδο 2007-2013, 71,5 δις δηλαδή, αντί για 78 δις κονδύλι που έχει στη διάθεσή του το ΕΚΤ. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί αυτή τη μείωση. Ποια είναι η λογική να έχουμε ένα κονδύλι που αντιστοιχεί και στις προσδοκίες του ΕΚΤ. Είναι ότι η κατάσταση που βιώνουμε είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο βιώνουμε μια βαθύτατη κρίση και διαρκώς αυξάνονται και τα αιτήματα που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αντίθετα τα κονδύλια μείωνονται. Υποτίθεται ένας από τους στόχους του ΕΚΤ είναι να υποστηρίξει την στρατηγική 2020, την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση, την πρωτοβουλία για τους νέους, την κινητικότητα στα πλαίσια του ΙΟΡΕΣ και να αντιμετωπίσει και τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει τα κονδύλια να είναι ανάλογα προς τις προκλήσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπίσει το ΕΚΤ. Για την πρωτοβουλία των νέων είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουμε ένα κατόφλι 25% για την ανεργία των νέων και η ηλικιακή ψαλίδα να είναι από τα 15 έως τα 24 χρόνια, ούτως ώστε να λάβουμε υπόψη τα περιορισμένα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας. Και για να έχουμε το αποτέλεσμα που περιμένουμε, ε, περιορίσαμε την ηλικιακή ψαλίδα. Ζητώ συγγνώμη, έσβησε το μικρόφωνο. Πανέρχομαι στην ηλικιακή ομάδα. 15 24. Αυτό προβλέπεται στην εγγύηση για τους νέους. Και εκεί είναι η πλειοψηφία των νέων που πρέπει να βοηθήσουμε Η ψαλίδα 24 έως 30 έτη έχει όντως υψηλή ανεργία, αλλά Η πλειοψηφία των νέων βρίσκεται στην πρώτη ψαλίδα. Η πρόορη εκταμίευση, το front loading, για το 2014 και 2015 έχει προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε αυτή τη διετία μπορούμε να υπερβούμε το κονδύλι της πενταετίας. 6 εκατομμύρια πάντως το αναγνωρίζουμε, δεν είναι πολλά λεφτά. Και το ΕΚΤ πρέπει να φέρει σε πέρα στους στόχους του. Ευχαριστούμε, συγγετής. Να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, λάβαμε, είχαμε πάντα λάβει υπόψη τον τελικό στόχο. Προτιμώ όμως να χάσω τώρα μια μικρή μάχη και όχι τον πόλεμο. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε στον πόλεμο. Όπως είπε και η Πρόεδρος, το Συμβούλιο ήδη έκανε πολλές παραχωρήσεις. Εν τέλει, δέχτηκε μια σειρά προτασιών μας, παρότι αντιστάθηκε επί μακρόν. Και μην ξεχνάτε ότι περιλαμβάνουμε στο κείμενο μια σειρά προϋποθέσεων πολύ πιο αυστηρών από την παλαιά περίοδο προγραμματισμού. Μην ξεχνάτε επίσης ότι και στον τομέα των συμφωνιών σύνδεσης θα έχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερο περιθώριο χειρισμού η Επιτροπή, κάτι που εξασφαλίζει ότι το κοινωνικό ταμείο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για πιο σημαντικούς στόχους, όπως την ανεργία των νέων ή άλλους στόχους. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε, κυρία Μωράν Σαρτιέ. Δεν χρειάζεται τώρα να επέμβετε και πάλι, έτσι δεν είναι μπράβο. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο της μερίσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ όλους και θα αναβάλουμε το σημείο 16. Θα γίνει μετά την ψηφοφορία μας, αν συμφωνείτε. για να μην υπερβούμε το χρόνο που είχαμε προβλέψει αρχικά για την ε, ψηφοφορία. Σημείο 17. Θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες. του Άνταμ Κώσε για τις κοινέ διατάξεις ε, για το ΕΚΤ, για την κατάργηση του κανονισμού 1083 του 2006. Ψηφίζουμε, υπενθυμίζω, ότι μόνο για τα ε, άρθρα 84.3 και 84 εδάφιο 5 ε, θα ψηφίσουμε για τις τροπολογίες διότι έχουν ήδη γίνει δύο ψηφοφορίες στις 5 Ιουλίου και στις 23 Απριλίου. Άρθρο 84, παράγραφος 3. Τροπολογία υπαριθμών 1 το εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχή. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την πρώτη τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. 12 υπέρ, 28 κατά, 4 αποχές. Απορρίπτεται η πρώτη τροπολογία. Θα ψηφίσουμε την ε, δεύτερη τροπολογία σε Έτζιο Γκουτιέρες Πρίτο και την τρία της κυρίας Μογάν Σαχτιέ και την κυρίων Σρέντερ και Λάμπερτ. Προτείνω απευθείας να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Κάποιος από τους σοσιαλιστές προσπαθεί να μπερδέψει την κάλπη. Εντάξει, ρυθμίστηκε, πέρας. 32 υπέρ, 12 κατά. 7 απόχέ. εγκρίνεται. Άρθρο 84, παράγραφος 5. Συμβαστική Α. Από το Ελκ και, και τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Υπέρ της συμβαστικής α, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράρτημα 3, ακούατε. Η τροπολογία 6 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 6. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε για το σύνολο ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Tout le monde a Πέρας. 38 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια, κύριε Κόζα. Nous en venons au point 18. Euh, θα ψηφίσουμε για την ε, διαπραγματευτική ε, εντολή βάση του άρθρου 70 του ιστορικού κανονισμού για τις ε, επικουρικές συντάξεις και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων. Πρόκειται για διαπραγματευτική εντολή, ούτως ώστε ε, να καταλήξουμε σε συμφωνία στην αρχή της δεύτερης ε, ανάγνωσης. Χρειαζόμαστε 25 ψήφους ε, για να εγκριθεί η διαπραγματευτική εντολή και θα σας προτείνω δια της ηλεκτρονικής όδου να ψηφίσουμε. Παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, μία κατά, τρεις αποχές. Δίνεται η διαπραγματευτική εντολή και θα απαρτίζεται. απ. κύριε Έρη. Από ό,τι βλέπω, κάποιοι δεν έχουν τις κάρτες τους μαζί για να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Δεν πρέπει να το διερευνήσετε. Μα είδατε στο αποτέλεσμα ότι είχαμε 40 ψήφους υπέρ στην οθόνη και εγώ είπα 40 41. Γι' αυτό ακριβώς επειδή έλαβα υπόψη ε, ε, ότι δεν έχουν όλη την κάρτα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ριόμενε Ρόιτεν που εκπροσωπεί το ΕΛΚΕ, Νταχντά από τους σοσιαλιστές, ε, Χάρκιν Αλντελ, Λάμπερτ Πράσινη, Τσίμερ για την ΚΟΕ, Καμπνόχ για τους συντηρητικούς. Αυτή είναι η σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Δεκαεννέα. Πρόταση Οδηγία Συμβουλίου Κοινοβουλίου για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Είναι το σχέδιο γνωμοδότησης της Μαρή Κορνέλισεν θα καταθέσουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Γυναικών που είναι σε αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, η πρώτη συμβαστική υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Article 3. L'amendement 111, est un amendement... Ε, με την τροπολογία 11 ε, αντικαθιστούμε τον DB Ποιοι είναι οι πέντε τροπολογίας αυτής 111. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, θα ψηφίσουμε το DB τριών πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Όχι, καλά. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε ε, στο άρθρο 4, παράγραφος 1, συμβαστική ε, δύο πολιτικών υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίθηκε. Άρθρο 4, για συμβαστική ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ. πέρας. 22 υπέρ 19 κατά, όντως εγκρίθηκε. Μετά, συμβαστική ε α, δύο ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Ε α. Παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 23 προς 17 με 7 αποχές εγκρίνεται. Πάμε στους τίτλους. Τροπολογία 1 του, της ηγήτρας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 43. Μπλίνκεβιτς ούτε είναι συμβατή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Μινοντόρα κλειβέτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρα. Άρθρο 2, εδάφιο 1, η 108 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Για την 108. Παρακαλώ. Tout le monde Ψήφισαν όλοι, πέρασε. 24. ψήφοι υπέρ 18 κατά εγκρίθηκε όντω. Άρθρο 2.8, η 109 της Ευελίν Ρέγκνερ είχε απαλληφθεί μια αράδας, αλλά έχει καταπέσει και άρα δεν την ψηφίσουμε και θα περάσουμε στην 110 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Άρθρο 4 για τον τίτλο, τροπολογία 22 της εισηγήτριας υπέρ κατά άποχες επαλήθευση για την 22. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 24 προς 18 εγκρίνεται. Η 115 για το ίδιο θέμα, Γιούτα Στάινερο και Πέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά, ε, Σαρίε 121 είναι κατά εισηγήτρια υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, παράγραφος 2, 122 Ρέγνερ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 123 Μπλίνκεβιτσούτε είναι συμβατή, προτείνει αποχή εισηγήτρια υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 124 Γιούτα Στάινρουκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4, παράγραφος 3, 125 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 126 της κυρίας Ροντσούλη συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παραρθρό 4 παραγραφός 4 26 της συγκεκριτρίας της είναι υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 της κυρίας Βλυνκεβιτσούτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 εσάια κατά αποχές απορρίπτεται. 27 της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 παραγραφός 5 συμβαστική F από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκτη παράγραφος 28 της εισηγητρίας για διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 παράγραφος 7, 132 Μπλυνκεβιτσούτε, καταπίπτει. Όπως και 29 και 133. 5-1 συμβαστική G, Z, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται παράγραφος 5, 2 ε, άρθρο 5 Τροπολογία H εγκρίνεται. 5-3. Τροπολογία 32 32-3. σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα έως το Future Selection Procedures υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 ε, άρθρο 5 παραφούς 4 Ναι, ναι, κατάλαβα ότι τα λέω πολύ γρήγορα. Άρθρο 5, παράγραφος 4, 141, Βλυκεβιτσούτα. 151 της κυρίας Μπλοκεβιτσούτα. Ψηφίζονται μαζί. Συγγετρία είναι κατά. Υπέρ παρακαλούμε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5-4. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 6-2. Συμβαστική Ι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6-2-α α45 και διαγραφή υπέρ κατά αποχές απερίφθη 146 πλην και υπέρ κατά αποχές απερίφθη Επαλήθευση. 146. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 21 υπέρ. 20 κατά. Εγκρίνεται, είχατε δίκιο. Ε, αργήσατε. Article 6 Μετά το β' 39. 34 λέει η ομιλήτρια τη εισηγητρία. Ψηφίζουμε. Υπέρ του 34. Υπέρ. Κατά. αποχές απρίφθη 147 Λούτβινξον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 εισηγητρίας υπέρ κατά άποχες απερίφθη 36 της υπέρ κατά άποχες απερίφθη 37 της υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 148 εσαϊά υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7-1 συμβαστική J τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8-3 πρώτη υποπαράγραφος K συμβαστική δύο ομάδες υπέρ κατά αποχές απερίφθη και ψηφίζουμε την 154 Σάια, υπέρ κατά εποχές Εγκρίθηκε. Τριάντα εννέα. Υπέρ. Τριάντα εννέα της συγκεντρίας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. εκατόν πενήντα επαλήθευση της 39. Άρχεται η σοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 25 υπέρ 19 κατά η τροπολογία 152 εγκρίνεται και σημειώνω ότι λειτουργήσαν ικανοποιητικά όλα τα μηχανήματα χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση τεχνικού. Η 153 έχει αποσυρθεί, όπως και η τεταράκοντα, και μπορούμε να προχωρήσουμε στην 155 τροπολογία της εισηγητρίας με προφορική τροπολογία. Συμφωνούν οι πάντες με αυτήν και μπορούμε να ψηφίσουμε την 155. Λοιπόν, με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 9.1.156 Μπλίνκεβιτσούτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9.2 υποπαραγραφος πρώτη 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 εσάγια υπέρ κατά άποχες θα επαληθεύσουμε την 157 ψήφισαν οι πάντες πέρας δεν εγκρίνεται 9, 2, 2, 159, Μπλικεβιτσούτε υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ. αποχές εγκρίνεται. 160 συγγνωμη περ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 9-3 161 να επαληθεύσουμε την 160 Άρχιτε ψηφοφορία, ψήσατε όλοι υπέρ ψηφοφορία. 161 Λουτβίνξον υπέρ. Κατά. Αποχές. απερίφθη 162 ούτε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 163 Χάρτς Πέτερ Μάρτιν. Υπέρ. Κατά. αποχές Απεριφθεί. 9-4. 164 βιτσούτε για διαγραφή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10 τίτλος 165 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 166 Την ψηφίζουμε τώρα όμως. Την 64 την έχουμε ψηφίσει. Πρέπει να ψηφίσουμε και την 165. Α, όχι, μπορούμε. Υπέρ. Κατά. Σε 166. Αποχές εγκρίνεται. 167 Bauer υπέρ. Εγκρίνεται 166, δεν έχει αποσυρθεί και άρα μπορούμε να ψηφίσουμε την 167. Λέει στα αγγλικά τώρα η, ομιλήτρια. Κατά αποχές απερίφθη. Στα δεδομένου ότι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τη σκέψη. 45 της κυρίας Χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 της ιδίας υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 χάρκιν υπέρ κατά ο κύριος Έρη είναι λίγο ταραγμένο στην ώρα της ψηφοφορίας. Τον ενοχλείται και δεν μπορούμε να ψηφίζουμε. Άμα είναι να ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Αλλιώς θα διακόψουμε. 49 Χάρκιν υπέρ. Αποχέ εγκρίνεται. Αιτιολογική 8, τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 9, 51 Μπάουερ υπέρ κατά αποχέ απερίφθη. 52 Χάρκιν υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 53 ροντσούλι υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται φαντάζομαι, αλλά ας το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν πάντες. Πέρασε. υπέρ, 22 κατά δεν εγκρίνεται. 55 Χάνς Πέτερ Μάρτιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 56 Ροντσούλη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 14. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 Χάρκιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 65 συμβατή υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 16. 66 Μάρτιν υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 67 συμβατή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Στην αιτιολογική σκέψη καταπίπτουν τροπολογίες. Πάμε στην 70 Χάρκιν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εβδομήντα ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72. Καταπίπτει. Τροπολογία 9. Της συγκεκριές υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την 9 της συγκεντρίας. παρακαλώ. Άρχεται η ψηφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 16 υπέρ 29 κατά. Υπερευθυντική. 75. Λούτβιξον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22. Σεβαστική β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έντεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται 24 υπέρ, τροπολογία 12 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται 82 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα τεσσερών, ομάδων υπέρ κατά. Αποχή εγκρίνεται 85 της ηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86 της εισηγητίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές επερίφθη 87 καταπίπτει. 88 ούτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαεπτά διαγραφή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. mais donc, donc il faut. Excusez-moi, je me suis trompée entre 90 et Ζητώ συγγνώμη, μπέρδεψα το 90 και το 92. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και να ψηφίσουμε την τροπολογία. 91, Λούντβιξον. 91. Το δέχεται η συγκεκριά. Ευχαριστούμε. Ψηφίζουμε 31 Λούτβιξον υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται και ζητώ συγγνώμη από τον συντάκτη. 32, 18, της ηγετρίας υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90, αν ναι, επαληθεύσουμε τροπολογία 18, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν πάντε, πέρα φοφορία. 23 υπέρ, 22 κατά, είχατε δίκιο, εγκρίνεται. 33-95 Μπλίνκεβιτσούτε υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 19 της συγκητρίας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 Λούντβιξον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβατική 97 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική D δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εκατόν δύο βιτσούτε υπέρ Κατά. Αποχές. κατά 103 της ίδιας συντάκτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο άρχεται. Πέρας. 37 υπέρ, 5 κατά, 4 εποχές, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και όλους όσοι έλαβαν μέρος στην διαπραγμάτευση. Και σας καλούμε να δείξετε σθένος και παρησία εκπροσωπώντας τις θέσεις της Επιτροπής μας σε πραγματεύσει με τις κατ' ουσίαν αρμόδιες επιτροπές και τώρα περνάμε στο σημείο 20. Όπου ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης, όχι. Την έκθεση πρωτοβουλίας Σγκαμ, έκθεση πρωτοβουλίας για την ανεργία των νέων πιθανές λύσεις επί των οποίων επί έχουμε τρία σχέδια γνωμοδότησης από την Επιτροπή Πολιτισμού, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Γυναικών. Πριν την παράγραφο 1, τροπολογία 88 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 91 και 92 ταυτόσιμες του ίδιου συντάκτη. Κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 93 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται επίση. 94 σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Μέχρι τη λέξη The Affected Youth, υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Θα κάνουμε έλεγχο για το πρώτο τμήμα της 94. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 1. συμβαστική J. Κύριε Ρέγνερ, τι θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, μια προφορική τροπολογία θα ήθελα να καταθέσω στην συμβαστική ε, J με τη διατύπωση compensated internships, αμοιβόμενες ε, πρακτικές ασκήσεις και εγώ θα ήθελα με τη λέξη Fairness μπρος στο κείμενο, δηλαδή δίκαια αμοιβόμενες, ή σωστά αμοιβόμενες. Με την τροποποίηση αυτή ψηφίζουμε το J. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 102, της Μόνικα Παναγιώτοβα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103, Μέρφυ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105, Σέρκας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 ημίδη κιουρούνεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 1, συμβιβαστική K από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 116 χίος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όπως και 117 που είναι ίδια. 118-119. ίδιες ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Μετά την παράγραφο 1. Παράγραφο 9 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 της Επιτροπής Κιούλτ εν μέρη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Συμβαστική L τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2, 134, Παναγιώτοβα, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 137, Σέρκας, υπέρ, 137 είναι η τροπολογία σας. Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 McIntyre, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 Παναγιώτοβα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 Κλειβέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρα καταπίπτει η επόμενη της ίδιας συντάκτριας μετά την παράγραφο 2 ένα παράγραφος επιτροπή Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το, για το εμπλεκόμενο κομμάτι. πέντε της Επιτροπής Κιούλτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 παράγραφος της Επιτροπής Κιούλτ εν μέρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πέντε παράγραφος της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Επιτροπής υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 6 της Επιτροπής Ρέζη εν μέρη τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Συμβαστική M. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε. Ε, 145 qui est compatible, je le mets au... 155 που είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Διοθόνιο μιλείτε. Ποιοι είναι υπέρ. 145. Όχι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 145 που είναι συμβατή με την M. Ποιοι είναι υπέρ της 145. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα που ξεκαθαρίσαμε γιατί ψηφίζουμε. Μετά την παράγραφο 3, 149, Ρέγνερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 150, Είναι Κριστίνα Ζούπερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, 153 τροπολογία. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Στην παράγραφο 4, συμβαστική N, τεσσάρων ομάδων. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Άρα 168 τροπολογία μετά την παράγραφο 4. Υπέρ εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, 21, εν μέρη της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24, της Επιτροπής Κιούλτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά α... Τι κάνουν εκεί οι φιλελεύθεροι να κάνουμε έλεγχο για την, επιτροπή, για την τροπολογία 8 της Επιτροπής Γυναικών να έχει την ψηφοφορία. Κάποιος ΕΛΚ ψήφισε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δύο. Πάντα υπεράριθμοι ή του ΕΛΚ. Κάντε μια μικρή προσπάθεια. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορία. 26 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 20 επιτροπής γυναικών υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 5. 171 του Πολ Μέρφυ που είναι καταργητική. Υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική όμικρον. Ο εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 5, 180 τροπολογία σε δύο τμήματα κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα χωρίς την λέξη as well as putting υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιο είναι υπέρ της προσήκης της πρότασης που αναφέραμε, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 5, 181 της Αντιπρόεδρου Ζούμπερ και του κ. Πολ Μέρφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 του Χάιντς Μπέικερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 σε δύο τμήματα μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα χωρίς το social security benefits all their interns. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με την προσθήκη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 5, 193 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, συμβιβαστική πι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6. 202 τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. 103 ε, λέει ο μιλήτρια, 203. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 κουπάκης υπέρ κατά αποχές δεκτή. 206 τυρίνεν Κρίστενσεν υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Η 207 που πάκης μπορεί να γίνει να ψηφθεί υπέρ, κατά. Δεν ψηφίζει. 207 υπέρ, κατά αποχές η 207 εγκρίνεται με τη θετική συνεισφορά των απεχόντων. Μετά την παράγραφο 6, παράγραφο 7 της Επιτροπής Γυναικών, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 7, συμβιβαστική Q, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 7, Μετά την παράγραφο 7, 220 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 7 Παράγραφος 17 της Επιτροπής Πολιτισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Συμβαστική ΆΡΜ, Δύο ομάδων. Υπέρ κατά. Αποχές. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο ή να πούμε ότι εγκρίθηκε. Έλεγχος για, το για τη συμβαστική άρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι είναι πολύ από το ΕΛΚ. Ως ήθιστε σήμερα. Διορθώθηκε η κατάσταση. Πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ 17 κατά 4 εποχές εγκρίθηκε. Μετά την παραγραφό 8. 230 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για 230. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 22 υπέρ. 24 κατά. Όντως απολύφθηκε. Παράγραφος 5 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 της ίδιας Επιτροπής υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εν μέρη η παράγραφος 18 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 9. Συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ κατά υπέρ της 236. Υπέρ. Υπέρ της 236. Κατά. Αποχές. Πέρασε. Παράγραφος 10. Συμβιβαστική τι τριών ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 249, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 250, τσούμπερ, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 12 παράγραφος Επιτροπής Πολιτισμού, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 14 της ίδιας επιτροπής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 11, συμβιβαστική U, τεσσάρων, τριών ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Μετά την παράγραφο 11, συμβαστική UU, τεσσάρων ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Συμβιβαστική Β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 13. Συμβαστική W. Υπέρ. Λάθος, λάθος. Λάθος, λάθος μου. Με ακούλπα. Μετά την παράγραφο 12. Μπορούμε να ψηφίσουμε εν μέρη την 127, ε, 277 διορθώνει η ομιλήτρια. Μετά την παράγραφο 12. Κατα, για ένα τμήμα της 277 ψηφίζουμε. Πολλών συντακτών που δεν θα διαβάσω, τον οποίο τα νόματα δεν θα διαβάσω. Αλλά είναι η κυρία Ρομπέρτα Αντζελίλη μεταξύ αυτών. Και η συγκίτρια είναι υπέρ. Δεν ξέρω τι, τι άποψη έχουν οι σοσιαλιστές. Ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα για την 277. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ίδια κατάσταση για την 278 για το τμήμα που μας αφορά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 21 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 της ίδιας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 της Επιτροπής ρέζει εν μέρη μόνο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Συμβιβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά τη 14, 298 τροπολογία, υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 299 υπέρ κατά αποχές, δεκτή. Στην παράγραφο 15, συμβαστική Y, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 19 της Επιτροπής Κιούλτ, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 16, συμβιβαστική Z, 5 ομάδων, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για την παράγραφο 47. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 17. Amendement 318 de Madame. 318 Steinbrück κατά δύο, σε δύο τμήματα μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα, χωρίς τη λέξη stress the need. Όχι, το πρώτο μέρος, το πρώτο, stress the need μέχρι of their traineeship. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παραγραφή 17, τροπολογία 319 Τσούμπερ Μέρφυ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά τη 17 τροπολογία 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για 321. Ψηφίσαμε πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ 18 κατά. Ευχαριστώ για την επαλήθευση. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 25 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 26 της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18 συμβιβαστική ΒΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 18 τροπολογία 324 και 26 ταυτόσημες. Ψηφίζουμε μαζί και τις δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 325 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 327 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 328 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 329 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 330 Έχω καλά νέα. Μετά από έρευνα την 330 μπορούμε να την ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κακά νέα για τους συντάκτες της τροπολογίας. 331. Κατέπεσε. Παράγραφος 3. Ως προσεσμένος αφορά της Επιτροπής Ρέζι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 4 Επιτροπή Γυναικών υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 6 γυναικών υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Εν μέρη 9 τη Επιτροπή Γυναικών υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 11 γυναικών υπέρ, κατά αποχές θα γίνει έλεγχος τη παραγράφου 11, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε τη ψηφοφορία. 19 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. 12 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 16 τη ίδια επιτροπή υπέρ, κατά, απόχε, εγκρίνεται. 17 τη ίδια επιτροπή υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 18 της ίδιας επιτροπής. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 της ίδιας επιτροπής. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προχωρούμε στα σκεπτικά. Ένα κόζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 της ίδιας υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 της ίδιας υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 χείρος υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τσεκ. Έλεγχος. Για το 12. Άρχεται ψηφοφορία. Ένας του ΕΛΚ παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 20 κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη α, η α παραγωγή των γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εν μέρη η β της ίδιας επιτροπής υπέρ κατά αποχές έλεγχος για, την, το αντίστοιχο τμήμα της παραγράφου β τη Επιτροπή Γυναικών. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε. Πέρα ψηφοφορία. Πάλι ένα του ΕΛΚ παραπάνω. Πέρα ψηφοφορία. 20 υπέρ 21 ψήφοι κατά. Δεν εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Γ μετά το Β. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη C. Συμβιβαστική δέλτα τριών ομάδων υπέρ κατά απόχέ, δεκτή. Μετά την αιτιολογική σε τροπολογία 32 Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την αιτιολογική σε συμβιβαστική FF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σε τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 34. Άρχιδη ψηφοφορία. Πάλι στο ΕΛΚ πολύ πολύ. Επιμένει το ΕΛΚ. Επιμένει ακόμα. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 25 κατά. Δεν περνάει το 34. Το 35. Ρέγνερ. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Στην αιτιολογική ντε συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά από την αιτιολογική ντε τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μπορούμε να ψηφίσουμε. πέντε μπορεί να ψηφιστεί υπέρ κατά αποχές. Αν σηκώνετε τα χέρια σας, μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί τις 45 ποιοι είναι υπέρ. δεν καλύπτεται η 39 από τη συμβαστική. Έπεφτε, θα, κατέπεφτε, θα κατέπεπτε η 45 μόνο αν είχε εγκριθεί 39. Επειδή δεν ψηφίσαμε χωριστά την 39, μπορούμε να ψηφίσουμε τη 45. Το θέμα είναι τι λέτε εσείς. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 21 κατά, 4 αποχές. Δεν εγκρίνει 45. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την αιτιολογική δέλτα, συμβαστική F των υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική δέλτα, δύο τροπολογίες οι ίδιες. Η 48 και η 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 στην αιτιολογική σκέψη ε υπέρ κατά αποχές Υπέρ της 51. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52. Σύμβατη υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 56 Ρέγνερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58. Νομίζω ότι ψηφίζεται. Ψηφίζουμε την 48 ε, γιατί απορρίφθηκε το 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική F, συμβαστική G, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το F, 66 τοπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην αιτιολογητή G, συμβαστική H, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική G, συμβαστική I, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική G, τοπολογία 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 απολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα αντίστοιχα τμήματα της 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85-86 οι όμοιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται το αντίστοιχο τμήμα της παραγράφου Δέλτα της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται G της ίδιας επιτοπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H της ίδιας επιτοπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος J της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σ της Επιτροπής Γυναικών υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. F της ίδιας Επιτροπής υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. G της ίδιας Επιτροπής υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. H της ίδιας Επιτροπής υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. έλεγχος για την AIDS της Επιτροπής Γυναικών Άρχεται ψηφοφορία. Το ΕΛΚ συνεχίζει την τακτική του. Υποχώρησε. Μπορεί, πήρε περισσότερες, τώρα ξαναβάλετε μια κάρτα, αν θέλετε. Πέρα, ψηφίστε το όλοι πέρα τη Ένα με τέσσερις αποχές. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο. Το αντίστοιχο τμήμα της παραγράφου I της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. J της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κ. της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το αντίστοιχο τμήμα της L της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. N της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε ολόκληρη την έκθεση. Όχι. Κύριε Σέρκας. Μπορείτε να ελέγξετε αν μετά την 11 παράγραφος η 264 κλειβέτη ψηφίστηκε, μπορείτε να το τσεκάρετε. Μετά την 11, 264 τροπολογία. Έχετε δίκιο. Δεν την ψηφίσα. Στη σελίδα 19 λοιπόν, στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Μετά την 11η παράγραφο, και την συμβαστική UU 264 της κυρίας Κλιμέτση. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονική επαλήθευση, ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν του συνόλου. Άρχεται η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ υπεράριθμο. Ψήφισαν οι πάντε Πέρα, Πέρασε 37 υπέρ. Μία ψηφο κατά. 7 αποχε και συγχαρητήρια κυρία εισηγήτρια. plastique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 Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε διάλειμμα. Δεν κάνουμε διάλειμμα. Παρακαλώ, καθίστε. Έχουμε πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά μπροστά μας. Doesn't work. They are all already in the summer break. yeah, yeah. I could see that. αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο σεβασμό για αυτούς που θέλουν ακόμη να δουλέψουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. It's incredible. Ah. Chut. Bien. Alors, euh, comme... Δεν θα μπορέσει να έρθει η κυρία Λόπε Φοντανιέ. Αντίθετα από αυτό που είχα πει πριν τις ψηφοφορίες και έτσι δεν θα μπορέσει να έρθει το απόγευμα κυρία Φοντανιέ. Άρα να ακούσουμε τώρα τι έχει να μας πει για το σχέδιο χρονομοδότησης στην έκθεση της Επιτροπής των Οικονομικών για το Ευρωπαϊκό Ξέμινο για το Στονισμό των Οικονομικών Πολιτικών Υλοποίηση των Προτεραιότητων για το 2013. Ησυχία, παρακαλούμε. Και την κυρία Λάμπερτ, θα τη δούμε το απόγευμα. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ που ε, δεν καθυστερήσα το θέμα αυτό. Ξεκινούμε σήμερα το διάλογο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και την εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013. Η αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας είναι η Οικονομική Επιτροπή για τα θέματα απασχόληση ωστόσο και βάσει του άρθρου 50 έχουμε αρμοδιότητα για θέματα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα και απασχόληση. Ελπίζω με την υποστήριξη και τη συμβολή όλων σας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα κείμενο που συμβαδίζει με τις αναγκαίες με τις υφιστάμενες ανάγκες όπως κάναμε και για την έκθεση της οποίας ήμουν συγγήτρια για τις μελέτες και τις προοπτικές για την ανάπτυξη για το 2013. Είναι προφανές, το είπαμε πολλές φορές στην Επιτροπή, ότι τα με οικονομικά μέτρα και τα μέτρα απασχόλησης είναι συμπληρωματικά. Οι κοινωνικές δε διαστάσεις δεν μπορούν να παραμείνουν υποκείμενες σε οικονομικά ζητήματα και μόνο. Είναι πολύ σημαντικό να προασπίζουμε τις κοινωνικές διαστάσεις στην έκθεση αυτή. Ο χρόνος που πρέπει να γίνει, μέσα στον οποίο πρέπει να γίνει το έργο είναι περιορισμένος. Έχουμε τις διακοπές του Αυγούστου και πρέπει να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να υιοθετήσουμε τη γνωμοδότηση αυτή στην συνάντηση της Επιτροπής μας 18 Σεπτεμβρίου. Ήδη είμαστε συνηθισμένοι στο να τρέχουμε πάντως και ελπίζω ότι παρά τις πιέσεις με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων θα καταφέρουμε έγκαιρα να το πετύχουμε. Είμαι αισιόδοξη πάντως. Το κάναμε και στην προηγούμενη έκθεση που ανέφερα. Στο προτινόμενο κείμενο επικεντρωνόμαστε στα θέματα που θεωρώ σημαντικά και, όπου, και που θα περιγράψω εντάχει. Πρώτον, θέλουμε να χτυπήσουμε την ανεργία ιδίω των νέων. Πρόκειται για μια προτεραιότητα της Ευρώπης πια, αλλά σίγουρα με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat του Μαΐου, η ανεργία, το ποσοστό ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,9%. 26 εκατομμύρια άτομα δηλαδή χωρίς δουλειά, από τα οποία 5,5 είναι νέοι. 23% στο, στην ομάδα του πληθυσμού. Στη χώρα μου δυστυχώ το ποσοστό αυτό είναι 50%. Στο Συμβούλιο του Ιουνίου τέθηκαν οι βάσει για την αντιμετώπιση τη ανεργία των νέων ω προτεραιότητα. Είναι αναγκαίο τόσο τα μέτρα που έχουν ε, προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στην πράξη. Θεωρούμε θετικό τη χρήση των διαθροτικών πόρων και όχι μόνο του, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά και την εφαρμογή στον, ε, στον αναπρογραμματισμό ε, πόρων που δεν έχουν δαπανηθεί. Επίσης θεωρούμε ότι τα έξι δις που θα δοθούν για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων να ενεργοποιηθούν αμέσως. Άλλο σημαντικό θέμα που σχολιάσαμε συχνά είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Είναι το ξεκίνημα για να ε, μπορέσουν οι νέοι να αντιμετωπίσουν τον ε, κόσμο της αγοράς εργασίας με καλές προοπτικές. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακάλυπτες λόγω διαφοροποίησης της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και ικανοτήτων. Γι' αυτό είναι αναγκαίο τα κράτη-μέλη να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να προσαρμόσουν τα προσόντα στην πραγματική ανάγκη της αγοράς. Άλλο θέμα σημαντικό είναι οι, άνεργοι, οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Τα κράτη-μέλη πρέπει να, επι, να ενισχύσουν την δυνατότητα επιστροφής των ατόμων αυτών στην αγορά με προγράμματα επανένταξης στην αγορά εργασίας ή ενδεδειγμένων συστημάτων ε, παροχών θα σχολιάσω εντάχει το θέμα των γυναικών. Οι γυναίκες είναι υπεύθυνε για την μέρη των παιδιών και των εξαρτημένων μελών της οικογένειας, γι' αυτό πρέπει να τις βοηθήσουμε να ξαναμπούν στην αγορά εργασία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σωστές υποδομές προστασίας ε, βρεφονιπιακών σταθμών και προστασίας ηλικιωμένων τα άτομα με αναπηρίες είναι προτεραιότητα για να μπορέσουν να υποστηριχθούν και να ενταχθούν στον χώρο εργασίας. Και εδώ είναι σημαντική η μόνιμη κατάρτιση που ανέφερα προηγουμένως. Κλείνω με το θέμα της αύξησης της φτώχειας. Η κρίση οδήγησε σε αύξηση της φτώχειας και του αποκλεισμού μεταξύ αυτών τη φτώχεια των παιδιών και τη φτώχεια των ανέργων. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν συστήματα κοινωνικής προστασίας που θα επηρεάζουν πραγματικά τους εμπλεκόμενους. Μια τελευταία παρατήρηση. Μιλήσαμε με την κοινωνία των πολιτών και τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι πρέπει να υποστηρίξουν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Φέτος πολλές χώρες, πολλά κράτη-μέλη, κατέβαλαν σχετική προσπάθεια. Ελπίζω η προσπάθεια αυτή να συνεχίζεται χρόνο με το χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σέρτζο Γκουτιέρες Ριώτο και μετά Κορνέλισεν και κανείς άλλος. Κύριε Κουτιέρες. Ευχαριστώ. Πρώτον, να εκφράσω την αναγνώριση μου για τη δουλειά της κυρίας ε, Λόπε Φοντανία και στη διαδικασία αυτή και συνέχεια και τη βούληση να τα βρει με όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Η καλή συμφωνία είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο έχουμε μια καλή σύμβαση, μια καλή συμφωνία για το κείμενο που πέρασε και το Φεβράριο με πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι το, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θέσουμε σαν ερώτηση, σαν ερώτημα σε, αυτό, σε αυτή την πρώτη έκθεση είναι τι από αυτά που αποφασίσαμε το Φεβρουαρίο τα πήρε η Επιτροπή και τα έκανε συστάσεις. Η απάντηση δυστυχώ είναι σχεδόν τίποτα. Πιστεύω λοιπόν ότι στην έκθεσή σας αυτή θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο κριτικοί σε σχέση με την προγενέστερη ε, κατάσταση για να είμαστε συνεπείς με αυτά που λέμε, για να πούμε στην Επιτροπή ότι ε, αυτό δεν μπορεί να κρατήσει και για να ε, μπορέσουμε να επιτρέψουμε να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Η στρατηγική που μας οδήγησε στο να συνεχίζει η Ευρώπη να είναι η μόνη περιοχή του κόσμου που συνεχίζει η αύξηση της ανεργίας, όπου οι χώρες πέφτουν σε μια βαθιά ύφεση και οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών, ιδίως φορά και Νότου, αυξάνονται ή να μειώνονται, θα έπρεπε να μας οδηγήσουν στο να είμαστε κριτικοί στην έκθεση αυτή και να απαιτήσουμε να προχωρήσει αυτό που εμείς ζητήσαμε το Φεβρουάριο. Και θέλω να τονίσω τρία πράγματα. Πρώτον, δεν μπορεί να είμαστε ανεκτικοί σε σχέση με τις προτάσεις που γίνονται για την αγορά εργασίας. Πρώτον, διότι η Επιτροπή κάνει ασυμμετρικές ε, προβλέψεις. Υπάρχουν δύο περιοχές στην Ευρώπη τελείως ασυμμετρικές και ως προς την προστασία των εργαζομένων και ως προς την μισθολογική δυνατότητά τους. Η Κομισιόν ακολουθεί μια στρατηγική η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της Ένωσης, αγνοώντας ωστόσο ότι ένα κομμάτι της Ευρώπης, ο Νότος ιδιαίτερα, πρέπει να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγικότητας, ιδίως το μισθολογικό. Κάτι που είναι εξαιρετικά ανητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εργαζόμενους. Με ανησυχεί το ότι δύο χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εκατομμύρια εργαζόμενοι έχασαν την προστασία των συλλογικών συμβάσεων. Και η Κομισιόν στις συστάσεις της ζητάει όλο και περισσότερες προσπάθειες. Δεν, δεν νομίζω ότι οι χώρες ε, ε, ζητώντας την αύξηση των, ε, της ε, ε, ανεργίας χωρίς καμία επίπτωση. Με ανησυχεί επίσης το copy-paste που έκαναν στο θέμα των συντάξεων. Εγώ είπα ότι η Επιτροπή πρέπει να ασχολείται με το θέμα τα βιωσιμότητας των ατόμων. Δεν μπορώ να καταλάβω ωστόσο ότι η Ένωση ε, πρέπει να επηρεάζει ε, και να αποφασίζει για την νόμιμη ε, ηλικία συνταξιοδότηση, για τα κριτήρια βιωσιμότητας, για τα κριτήρια άθρησης των, συντάξεων. Δεν νομίζω ότι μπορεί να, να δώσει κοινό παρονομαστή ούτε συμφωνώ να με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ενεργείας των νέων. Προφανώς το θέμα της εγγύησης των νέων δεν μπορεί να χαθεί Καλά λέει, συμφωνώ με το ότι είναι μια καλό, ένα καλό ξεκίνημα, αλλά έχουμε πολύ μεγαλύτερα ποσά μέσα, 20 δις ευρώ που πρέπει να ζητήσουμε. Όταν η επιτοπή και το Συμβούλιο φαίνεται ότι είναι θετικές στο να προκαταβληθούν τα δύο δις το πρώτα δύο χρόνια, θα έπρεπε να ζητήσουμε το τριπλά όπως ζητάει και το Παγκόσμιο Γραφείο Εργασίας. Τελευταία παρατήρηση. Μήπως θα θέλετε να τελειώσετε συνάδελφε. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Πρέπει επίσης να κατακρίνουμε την δημοκρατική διαδικασία. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει θέση τον Οκτώβριο για κάτι που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο από τα κράτη-μέλη. Αυτό μας γελιοποιεί. Δεν μπορεί το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να παραμείνει έτσι. Θα πρέπει να τηρήσει την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση της, ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Κορνέλσεν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχουμε καθυστερήσει πολύ και παρακαλώ να είστε σύντομοι. Βεβαίως, Καταρχάς ευχαριστώ τον την ε, εισηγητρία για την πρότασή της, η οποία αποτελεί μια καλή βάση. Έχουμε τη δυνατότητα φέτος με την ε, ε, ικανή ηγεσία της κυρίας Λόπε Φοντανιά για άλλη μια φορά να έχουμε μια καλή ε, γνωμοδότηση. Η Επιτροπή των Οικονομικών ίσως να έχει λιγότερο, λιγότερη σύμπνοια να εκδηλώσει στο εσωτερικό της και εμείς μπορούμε να περιμένουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε εκ τούτου για την Ολομέλεια. Τέσσερις παρατηρήσεις. Θα πρέπει να είμαστε πιο απερίφραστες προς τα θέματα της ε, δημοκρατίας θα πρέπει να μιλάμε πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή, ε, ήδη είχαμε δει ότι δεν θέλουμε η οικονομική διακυβέρνηση να αναπτυχθεί χωρίς πλήρη ε, εμπλοκή στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε επαναλάβει ότι επανειλημμένως Κάποιες φωνές λένε πως δεν υπάρχει δυνατότητα υπό τις συνθήκες, υπό την ισχύουσα συνθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να αναλάβει ρόλο στην οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό όμως δεν ισχύει. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια διοργανική συμφωνία για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ετήσια έκθεση ανάπτυξης και στις ε, έρευνες, στις μελέτες, εκθέσεις Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Δεν πρέπει επίσης να σιωπήσουμε ως προς τα θέματα των δημοσιονομικών συστάσεων. Οι καθυστερήσει για τα υπερβολικά ελλείμματα δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά. Η ανεργία των νέων επίση, ε, που ζητούμε πάρα πολύ θα πρέπει να συζητηθεί στι πραγματικέ διαστάσεις και αιτίε σχετίζεται με τη γενική ανεργία και την απουσία θέσεων εργασία σε ορισμένες περιφέρειες, περιοχές. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει η ε, χρηματοδότηση της ανεργίας των νέων να αποκλειστεί από τον υπολογιστό του υπερβολικού ελλείμματος για να δοθεί ευκαιρία για ε, νέες επενδύσεις και επίσης εν τέλει θα πρέπει να φροντίσουμε το θέμα των, ε, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας από τα κράτη-μέλη στις ε, περιοχές που παρουσιάζουν φαινόμενα ανεργίας. Ε, δυστυχώς και παρότι το έχει υποστήριξει και ο Επίτροπος Άνδρος, δεν έχουμε λάβει ακόμα, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτε το συγκεκριμένο. Κυρία Λόπες Φοντανέ, εγώ συμφωνώ απολύτως με τα όσα υπόθηκαν, δεν χρειάζεται να παρέμβω. Θα κάνουμε καλή δουλειά πιστεύω και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ και χαίρομαι. Ευχαριστώ την συγγήτρια. Τώρα, με πολύ στενά χρονικά όρια, 17 Ιουλίου ορίζουμε την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, 12 το μεσημέρι. Εξετάζουμε στις 5 Σεπτεμβρίου τις συμβαστικές της 18 και τις ψηφίζουμε την ίδια μέρα, γιατί 30 Σεπτεμβρίου ε, γκρίνει την εκθεσή της η Επιτροπή των Οικονομικών. Έχουμε κλείσει λοιπόν και το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Τώρα στο 23. Προτείνω να ξεκινήσει η ακρόαση. δημόσια ακρόαση με θέμα κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ένα ευρωπαϊκό σύστημα παροχών ανεργίας και τι θα μπορούσε αυτό να προσφέρει. Καλό λοιπόν τους εμπειρογνώμονες να έρθουν στο βήμα. avons Λοιπόν, πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται δημόσια ακρόαση για το ζήτημα αυτό που αποτελεί και ουσιοδέστατο επίκεντρο της συζήτησης ως προς την ε, θέσπιση μιας οικονομικής και νομισματικής ε, ένωσης. Έχουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες μεταξύ μας και τους ευχαριστώ που δέχτηκαν την ε, πρόσκλησή μας πέραν των εγγράφων τους έχετε και το έγγραφο του κυρίου Αρτ Τεμπούς από το ε, Ινστιτούτο Μπέρτελσμαν ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει ενώ ήταν προσκεκλημένος αλλά σας στέλνει γραπτά την τοποθέτησή του. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Γκέορκ Φίσερ πρώτο τον οποίο γνωρίζετε από καιρό, θα απαντήσει στις δύο ερωτήσεις που έχουμε θέσει. Ε, πρώτη ερώτηση, γιατί πρέπει να γίνει συζήτηση για το θέμα αυτό και δεύτερον, πώς. Γεώργ Φίσερ. Έχετε μακρά διαδρομία και γνώση στον τομέα αυτών μετά το Αυστριακό Υπουργείο Οικονομικών και Απασχόλησης, ε, γιατί είχατε διπλή ε, καθήκοντα, ήρθατε στην Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων το 1993 και ασχολείστε με την, με την κοινωνική διάσταση των εξωτερικών σχέσεων. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους. Με εντυπωσιάζει το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το θάρρο να θέσει αυτό το σημαντικό θέμα. Πρόκειται για έναν από του μακροπρόθεσμου ε, στόχου μα, αλλά πάντω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπω ξέρετε, ο κύριο Άντορ, ο επίτροπό μου, στου πρόσφατου μήνε έχει πολλέ φορέ επισημάνει το ζήτημα και προβάλλει το ζήτημα της Ευρωπαϊκής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και το σταθεροποιητικό παράγοντα που μπορεί να δραματίσει μια οικονομική διακυβέρνηση στον τομέα αυτό. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση σημειώνεται δε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει στήσει για άλλη μια φορά την ενίσχυση της οικονομικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Έχει ζητήσει επίσης καλύτερη επιτήρηση των ε, ε, κοινωνικών και εργατικών πτυχών και ένα πιο διεξοδικό ε, πρόγραμμα ε, για την ε, περιχαράκωση της οικονομίας και της απασχόλησης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και προβλημάτων ανεργίας και έχει στηθεί ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το ζήτημα των οικονομικών σταθεροποιητών για πρώτη φορά στο προσχέδιο για την ε, βαθιά αλλαγή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχει δε περιγράψει με την ιδέα μιας πλήρους ε, δημοσιονομικής επέκτασης της Ευρωπαϊκής Κοινωνισματικής Ένωσης και πιο ουσιαστική συνεργασία στα οικονομικά, γιατί βέβαια αυτά δύο ε, είναι αλληλένδετα. Επίσης, δε στο προσχέδιο αυτό, το blueprint, ε, επισημαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα λόγω της απουσίας των αυτοματών των σταθεροποιητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας έδωσα κάποιες διαφάνειες εδώ για να μπορέσω να εξηγήσω καλύτερα τα στοιχεία μου. Εγώ απλώς σας συνοψίζω προφορικά τα στοιχεία που βλέπετε αναλυτικά στις διαφάνειες. Σταθεροποιητής είναι εκείνο το πράγμα που όταν μια οικονομία ε, μπαίνει σε ύφεση και βλέπουμε να συρρυκνούται η οικονομία, το πορτοκαλί χρώμα που βλέπετε, εμφανίζεται με έναν αυτόματο σταθεροποιητή η δυνατότητα της διαφύλαξης ή της αυτόματης εμφάνισης των κοινωνικών ε, παροχών, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να ληφθεί αποφασία από κυβέρνηση ή από κοινοβούλιο, αυτομάτως τίθεται σε κίνηση ο μηχανισμός αυτός παροχής των κοινωνικών παροχών που ε, σε ένα βαθμό αντισταθμίζουν την υποβάθμιση στα εισοδήματα και ταυτόχρονα μειώνεται και η ε, φορολογία που επιβάλλεται, πληρώνει δηλαδή λιγότερο φόρο ο πολίτης. Βέβαια αυτό ταυτόχρονα ε, επιτρέπει να ενισχυθεί το εισόδημά του σε μια περίοδο ύφεση. Αυτό είναι λοιπόν ο αυτόματο σταθεροποιητή και κάτι άλλο που, όπως, που για κάποιον όπως, που όπως εγώ έχει δουλέψει σε οικονομικό υπουργείο ε, το θετικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να διαταράξουν τις οικονομικές δομές σε περίοδο ε, ανάπτυξης οικονομικής. Παραμένουν δηλαδή ε, περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασής τους. Και επίσης μακροπρόθεσμα με την ΩΝΕ ε, θα έχουμε να αναπτύξουμε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και μηχανισμούς. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιούμε το μηχάνημα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε πράγματα τα οποία ξέρετε πολύ καλά και εσείς. Την ανάπτυξη της ανεργίας στην Ευρώπη από το έτος 2000 και αυτό που βλέπετε ουσιαστικά εδώ είναι ότι για το πρώτο ήμιση της περίοδου, της περίοδου αυτής έχουμε βασικά μια σύγκληση στην ενεργεία, δυστυχώς προς τα άνω αρχικά, μετά προς τα κάτω, αλλά από το 2008 έχουμε μια πολύ σημαντική και ταχεία πόλωση στην ανεργία. Πρόκειται για μια περίοδο όπου θα μπορούσαν οι αυτοματοί να διαδραματίσουν πολύ χρήσιμο ρόλο, αν υπήρχαν. Για να δω πώς πάει αυτό μπροστά. Ε, εδώ. Και τι γίνεται λοιπόν όταν προχωρεί ταχαίως η ανεργία σε κάποιες περιοχές της Ένωσης. Εδώ έχουμε καταγράψει τις συνέπειες της δαπάνες για την κοινωνική πολιτική τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και διαπιστώνουμε ότι τα πρώτα χρόνια, βλέπετε το 2008 έως 2010, η κόκκινη γραμμή, μαζί με την υποβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας και οι δαπάνες ε, για τις κοινωνικές παραχές αυξάνονται, δηλαδή υπάρχει αυτός ο σταθεροποιητικός ρόλος. Μετά όμως η κοινωνική πρόνοια υποβαθμίζεται, μειώνεται πολύ πιο γρήγορα από τις σε προηγούμενες περιόδους ύφεσης, δηλαδή χάνει τον χαρακτήρα της ως ε, αυτόματου σταθεροποιητή και θα λέγαμε ότι τουναντίον επιδεινώνει την οικονομική ύφεση. Ε, πολλοί θα είναι λόγοι ασφαλώς, αλλά κάποιοι από αυτούς σχετίζονται με το ότι σε μια νομισματική ένωση τα κράτη-μέλη έχουν, έχουν χάσει ε, σε ένα βαθμό τη δυνατότητά τους, την εξουσία τους για αξιοποίηση των αυτόματων σταθεροποιητών. Σταματώ εδώ. Αυτό είναι ο λόγος πάντως για τον οποίο το θέμα αυτό το έχουμε φέρει στην επικαιρότητα και γι' αυτό ε, διατυπώνει αυτό το προσχέδιο προτάσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση λοιπόν, στην πρώτη σας ερώτηση. Γιατί το θέμα αυτό το έχουμε για συζήτηση. Σας προτείνω να κάνουμε το εξή ο καθένας να απαντήσει το πρώτο ερώτημα γιατί τίθεται έτσι ε, το θέμα προς το παρόν, δηλαδή Αυτό μου υπέδειξαν τουλάχιστον. Θα δώσω το λόγο στον Τωμά Φιλιππό ε, που έχει μακρά ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών στη Γαλλία. Σας δίνω το λόγο και πέντε λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε σε αυτό το πρώτο ερώτημα. Στα αγγλικά καλύτερα. Okay. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στη σημερινή ακρόαση. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Έχω πέντε λεπτά στη διάθεσή μου, μου είπατε. Ε, Είναι ευρύτερη η οπτική μου γωνία γιατί θα κάνω ένα παραλληλισμό με τη ΣΥΠΑ για να απαντήσω. Ταυτόχρονα δίνω και, ε, απηχώ την παρέμβαση του George Fisher ε, αυτή η έλλειψη αυτόματων σταθεροποιητών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν στη ΣΥΠΑ. Δείτε αυτή τη ε, τη γραφική συγγνώμη, παράσταση μέχρι το 2010. Ας πάρουμε πρώτα την φύση της κρίσης, που είναι μια κρίση χρέους, ιδιωτικού χρέους για την πρώτη τριετία. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες εδώ. Στον οριζόντιο άξονα βλέπετε τον αριθμό των οικοκυριών που δανείστηκαν ε, στην ανωδική φάση του κύκλου από το 2003 ως το 2007. Κάθε κουκίδα είναι μια πολιτεία τον ΗΠΑ ή ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί προσπαθούμε να συγκρίνουμε δύο μεγάλες νομισματικές ενώσεις. Κάτω δεξιά έχετε την Εβάντα και πάνω το Τέξας. Το μπλε τρίγωνο είναι η ΙΠΑ. Τα μέλη της Ευρωζώνης είναι με πράσινο χρώμα. D, Deutschland, Γερμανία, πάνω αριστερά. Την Ιρλανδία και την Ισπανία έχετε κάπου στη μέση, αν δεν κάνω λάθος. Τι βλέπετε λοιπόν εδώ. Στον οριζόντιο άξονα βλέπετε ε, στην ανωδική φάση του κύκλου πόσα ε, δανείστηκαν τα νοικοκυριά από το 2003 στο 2007. Ας πάρετε την Εβάντα γιατί είναι η πιο ακραία περίπτωση. Βλέπουμε ότι ο λόγος ε, του χρέους προς το εισόδημα ήταν 65 70%. Ε, και με τη μόχλευση φτάσαμε στο 170% για τα νοικοκυριά. Στο Τέξας δεν τροποποιήθηκε ο λόγος αυτός, ίσως 10%, ενώ στη Γερμανία ήταν μάλλον αντιντικός ο λόγος. Στον κάθετο άξονα βλέπετε τι συνέβη μετά, κατά τη διάρκεια της κρίσης και στις αλλαγές που σημειώθηκαν στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση. Ε, σε ποσοστιαίες μονάδες βλέπουμε τις αλλαγές ε, για την περίοδο 2007 ως το 2010. Σταματάω στο 2010, πρωτού αρχίσει η κρίση του δημοσίου χρέους. Βλέπετε πρώτα απ' όλα με ξεκάθαρο τρόπο ότι οι Αμερικανικές πολιτείες ή ε, τα κράτη της Ευρωζώνης που είχαν μεγάλη ύφεση και έχασαν πολλές θέσεις απασχόλησης είναι εκείνα που είχαν υπερμόχλευση για το ιδιωτικό χρέος. Ε, βλέπετε πόσο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση. Αυτό είναι στον πυρήνα της κρίσης. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Και αντίθετα με αυτά με τη λαϊκή θυμοσοφία, η απόκληση ήταν πολύ μεγαλύτερη στο ιστορικό των ΗΠΑ παρά στο ιστορικό της Ευρωζώνης. Ανάμεσα στο Τέξας και την Εβάντα βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη απόκληση σε σχέση με αυτό που βλέπουμε π.χ. ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία. Μεγάλες αποκλήσεις λοιπόν στη ΣΥΠΑ. Και έχουμε την εντύπωση ότι σε νομισματικό επίπεδο είναι σε βέλτιστο επίπεδο η ΕΠΑ. Ε, όχι λοιπόν, οι αποκλήσεις ήταν πολύ ευρύτερε σε σχέση με την Ευρωζώνη. Δεν χαρακτηριζόμαστε λοιπόν ε, ε, χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο μέτρησης ε, από μεγάλες αποκλήσεις όπως είπα. Στη συνέχεια βλέπουμε τη σχέση ανάμεσα στη μόχλευση και την κρίση, τη μεταγενέστερη κρίση. Δηλαδή με την απομόχλευση, περιορίζοντας και τη ζήτηση, βλέπουμε τη μείωση της ανεργίας. Όμως, οι δύο καμπύλε είναι σχεδόν πανομοιότυπες. Δεν μπορείτε με το μάτι να καταλάβετε ε, πού σημειώθηκε η πιο κατακόρυφη μείωση. Τι συμβαίνει αυτό ότι η απομόχλευση αναμονάδα χρέους ήταν ακριβώς η ίδια στη ΣΥΠΑ και στην ΕΕ. Αυτό μας εκπλήσει. Δηλαδή, ό,τι συνέβη, ο επιμερισμός του κινδύνου ήταν ε, παρομοιότυπος στις δύο αυτές νομισματικές ε, ζώνες. Αυτά το 2010 όταν ε, λειτουργούσαν αυτοί οι αυτόματοι σταθεροποιητές, όπως σας έδειξε και ο κύριος Φίσερ. Γι' αυτό έχουμε τους σταθεροποιητές διότι ε, σε, όταν σε δημοσιονομικό επίπεδο υπάρχει ένα περιθώριο μπορεί το κράτος να δώσει αυτόν τον αυτόματο σταθεροποιητή και είχαμε ε, ως προς τον επιμερισμό κινδύνου ε, εξίσου καλά αποτελέσματα όπως είπα αλλά ήταν καλύτερο το εφαλτήριό μας γιατί είχαμε μικρότερες αποκλήσεις ε, ε, και μικρότερο ιδιωτικό χρέος ήταν ε, για την περίοδο 2007-2010 μικρότερη η κρίση σε εμάς παρότι στη ΣΥΠΑ για να δούμε στη συνέχεια Αριστερά τώρα βλέπουμε τη ΣΥΠΑ και δεξιά την Ευρωζώνη. Έβαλα δύο γραμμές, την κόκκινη γραμμή για τη ΣΥΠΑ. Είναι ακριβώς η ίδια ε, καμπύλη που βλέπατε νωρίτερα. Και βλέπετε τι συμβαίνει ακριβώς στις ίδιες πολιτείες, αλλά στο δεύτερο ήμιση ε, της ε, κρίσης, δηλαδή από το 2010 ως το 2012. Βλέπετε ότι ε, λίγη η κρίση. Για αυτή τη διετία δεν υπάρχει πλέον αντίκτυπο, δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφορά προς την ανάπτυξη της απασχόληση σε σχέση με τη χαμηλή ή την υψηλή μόχλευση, ανάλογα με το αν στην πολιτεία υπήρχε υψηλή ή χαμηλή μόχλευση και βλέπουμε ότι είναι σχετικά θετική πορεία, αλλά έχουν συρρυκνωθεί αποκλήσει ανάμεσα στι Αμερικανικέ πολιτείε. Αν σταματήσετε τώρα εδώ και ζητήσετε από κάποιον από τον Άρη, ε, τι προβλέπετε για την Ευρωζώνη, ε, τι, θα είχε προβλέψει ότι θα ήταν λίγο καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με τι ΗΠΑ, ε, για αυτού του λόγου που προανέφερα. Όμω το αντίθετο συνέβη. Δείτε στη δεξιά πλευρά ότι έχουμε μεγάλε αποκλήσει ω προ την αύξηση τη ανεργία στην Ευρωζώνη και ε, έχουμε την μεταβλητή ε, στον κάθετο άξονα που το εξηγεί αυτό. Δεν είναι το ιδιωτικό χρέος πλέον. Είναι ε, το κατά πόσο οι κοινωνικές μεταφορές πιστώσεων αυξήθηκαν από τις κυβερνήσεις κατά την ανωδική φάση του κύκλου μιλάμε για προκυκλικά μέτρα ή υπερβολικές δαπάνες κατά την άνθηση της οικονομίας. Οι κυβερνήσεις που ξόδεψαν τα περισσότερα έπεσαν πάνω στον τοίχο και τη λάθος στιγμή έπρεπε να περικόψουν τις δαπάνες και δημιούργησαν αυτή την ε, βαθιά ύφεση. Ε, βλέποντας αυτό λοιπόν δεξιά, εγώ καταλαβαίνω ότι μετά το 2010 η έλλειψη ακριβώς επιμερισμού κινδύνου ε, επιδίνωσε σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, εμείς δημιουργήσαμε δηλαδή την κρίση. Αν είχαμε καλύτερα εργαλεία τόσο ώστε να μην μεταδίδεται η κρίση από το ένα κράτος στο άλλο, δεν θα είχαμε καταλήξει σε τόσο βαθιά κρίση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τους αυτόμους θεθεροποιητές και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε στον τρίτο ομιλητή, Φίσερ, είστε μέλος του DIV, του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών. Υπηρετήσατε στην ΕΚΤ και στην ΔΙΒ. Είστε ο κατεξοχήν εμπειρογνώμονας ε, που μπορεί να μας δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να έχω την, ε, το τηλεχειριστήριο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σας δείξω ένα σύστημα το οποίο έχουμε επεξεργαστεί μαζί με τον Σεμπαστίαν του Τζέιν από άλλο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ένα σύστημα αυτόματο σταθεροποιητή σε ένα, με, με ασφαλιστική κάλυψη ανεργίας. Θα ήθελα όμως να εξηγήσω πρώτα το γιατί χρειαζόμαστε μηχανισμό σταθεροποίηση στην ε, νομισματική ένωση. Θα είμαι σύντομος ε, όσο μπορώ και βεβαίως ε, στα όσα είπαν οι συνάδελφοι θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ, αλλά μια και προέρχομαι από την νομισματική περισσότερο πολιτική, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό. Η κοινή νομισματική πολιτική δεν μπορεί λοιπόν να λάβει υπόψη του γεγονός ότι δεν είναι συντονισμένη και είναι πολύ διαφορετική οι κύκλοι, οι οικονομικοί και ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση των περιοχών ή των χωρών εκείνων που έχουν ε, μεγάλη ανάπτυξη, ταυτόχρονα αυτό έχει επιπτώσει σημαντικές για τις χώρες οι οποίες παρουσιάζουν ε, ύφεση. Είναι το λεγόμενο Taylor Rules στα επιτόκια, επιτόκια τα οποία μπορεί μια κεντρική τράπεζα στηριζόμενη στο, σε μια κατάσταση κύκλου επιχειρησιακού, εγώ δεν βλέπω από εδώ βέβαια, αλλά ίσως να μπορείτε εσείς να το δείτε, ε, να το καλύψει. Βλέπετε λοιπόν ότι το επιτόκιο για την Ισπανία που είναι πολύ ψηλότερο στην περίοδο πριν από την παγκόσμια ύφεση, πριν το 2008 δηλαδή, και βλέπετε ότι το επιτόκιο για τις πιο αδύναμες χώρες, τη Γερμανία, Φερρυπίν, είναι αυτές που δηλαδή παρουσιάζουν το χαμηλότερο ε, επιτόκιο, είναι πολύ χαμηλότερο και μετά βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσανατολίστηκε σε ένα επιτόκιο που ανταποκρινόταν στις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών με το χαμηλότερο επιτόκιο και ως εκ τούτου οι χώρες οι οποίες είχαν μια σταθερή οικονομική κατάσταση και είχαν υψηλή ανάπτυξη όπως η Ισπανία και άλλες χώρες του Νότου υπερθερμάνθηκαν. Γιατί η νομισματική πολιτική ήταν για αυτές υπερβολικά χαλαρή. Σε μια οικονομική ένωση βέβαια το αντεπιχείρημα είναι ότι αν δεν υπάρχει ο σταθεροποιητής η νομισματική πολιτική χρησιμοποιείται η δημοσιονομική πολιτική ο σταθεροποιητής. Αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι, δηλαδή ε, σταθεροποιητές εισάγονται προκειμένου να ε, αντισταθμίσουν ή να αναλάβουν ακόμα και το ρόλο της νομισματικής πολιτικής ως σταθεροποιητή. Ωστόσο βλέπουμε ότι αυτό δεν δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε χώρες με πολύ μεγάλη διασύνδεση μεταξύ τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασύνδεση και εμπορική και αν ε, Ε, μέσω του εμπορίου διαχέεται κατά κάποιο τρόπο η ανάπτυξη γιατί μπορεί κανείς να πληρώνει τους φόρους στην ε, χώρα του αλλά διαχέεται το εισόδημα ε, σε άλλες χώρες λόγω της, οικονομικής, λόγω της εσωτερικής αγοράς. Ένα άλλο φαινόμενο που βλέπουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική έχει περιορισμένες δυνατότητες μέσα σε μια οικονομική ένωση. Όχι μόνο συντονισμό δημοσιονομικής πολιτικής μέσω του, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιορίζει την ευελιξία της οικονομικής ένωσης, αλλά ταυτόχρονα και οι ε, χρηματοπιστωτικές αγορές ε, πιέζουν τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων σε μια πολύ περιορισμένη δυνατότητα χρήσης της δημοσιονομικής πολιτικής ως μέσου. Γι' αυτό ήταν στην Οικονομική Ένωση πολύ περιορισμένη η δημοσιονομική πολιτική, γι' αυτό δεν μπόρεσε να δώσει α, α, α, αντιστάθμιση σε προβλήματα ε, διακύμανσης των ε, δικτών. Και από την άλλη έχουμε συστήματα δημοσιονομικά, τα οποία στόχο έχουν να αντισταθμίσουν τη σταθεροποίηση, την απουσία σταθεροποίηση της ε, οικονομικής πολιτικής και της δημοσιονομικής πολιτικής. Είναι ένα αυτόματο σταθεροποιητή μεταξύ ε, χωρών. Υπάρχουν αυτόματοι σταθεροποιητέ μέσα στι χώρε, φερειπίν μια ασφάλιση κατά τη ανεργία, με έναν αυτόματο σταθεροποιητή, που θα μπορούσε να εισαχθεί για όλε τι χώρε. Αυτόματε μεταφορέ δηλαδή μεταξύ των χωρών που βρίσκονται σε ανάπτυξη και εκείνων που θα στέλνουν τα χρήματα αυτόματα, τους σπόρους αυτούς, αυτόματα προς τις χώρες που αντιμετωπίσουν την ύφεση. Και έτσι η νομισματική πολιτική θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των ε, διακυμάνσεων της, ε, του οικονομικού κύκλου και βέβαια να συγκρατήσει έτσι την πτυτικότητα στην Νομισματική Ένωση. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Τελευταίος παρεμβαίνουν ο Μανουέλ Καλτέρα Καμπράλ. Σπουδάσατε και δουλέψατε ως δημοσιογράφος. Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών της Πορτογαλικής Κυβέρνησης, ενώ δουλέψατε και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Άρα, μπορείτε να απαντήσετε το πρώτο ερώτημα. Πού είναι το πρόβλημα και γιατί θέτουμε το ερώτημα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Δεν ήξερα τι προσέγγιση να ακολουθήσω. Προτίμησα την προσέγγιση των ασυμμετρικών σοκ. Διότι, ήταν, ε, μια, γιατί από εκεί προήρθε η ιδέα των αυτόματων σταθεροποιητών και που κάπου ξεχνάμε στη συζήτηση της, της κρίσης όταν εξετάζουμε το, τη σχέση της κρίσης ως ποσοστό του ΕΠ ξεχνάμε ότι ένα κομμάτι της ιστορίας είναι η αύξηση του χρέους, άλλο ήταν η αύξηση του ΑΕΠ και ειδικότερα η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Και χώρες που έχουν αύξηση ανάπτυξη ΑΕΠ έχουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή το ΑΕΠ ε, ε, αυξάνεται μόνο εγχώρια, όχι με εσωτερικές επενδύσεις, χωρίς να αντιμετωπίζονται εξωτερικές ανισορροπίες περισσότερες χώρες που έχουν προβλήματα. Κάτι που ξεκίνησε νωρίτερα με τα συμμετρικά σοκ πηγαίνουν λοιπόν στην ευθεία γραμμή των ε, βελτιστοποιήσεων ε, κάθε Όταν οι χώρες μπαίνουν σε, ενιαία, σε ενιαίο νόμισμα και χάνουν την ε, τη νομισματική αυτονομία τους, ε, εμφανίζουν άλλους τρόπους ε, βελτίωσης της καταστασής τους, δημοσιονομικοί κανόνες κλπ. Τα εργαλεία αυτά πρέπει να τα παρακαλύψει η χώρα σε μέσω πρόθεσμη προσαρμογή, ιδίω αν αυτή η προσαρμογή απαιτεί, είναι σύμμετρη, δηλαδή επηρεάζει διαφορετικέ ε, χώρε σε διαφορετικού τρόπου. Η, η βέλτιστη νομισματική πολιτική θα παίρνει διαφορετική από χώρα σε χώρα και αυτό δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο νομισματική Ένωση. Για να ελαχιστοποιήσουμε του κίνδυνου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό ήταν κομμάτι της ομιλίας, ε, του, του, της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί να υπάρχει κινητικότητα των παραγόντων στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης. Υπάρχει ήδη μετανάστευση από τον νότο στο βορρά ή και δικές μεταφορές σταθεροποιητών που σημαίνει ότι οι χώρες που έχουν καλύτερη κατάσταση μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια σε χώρες με μικρότερη, σε δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση που θα μπορούσαν να παράσχουν με άλλα λόγια ε, επιδόματα ανεργία χωρίς υπερβολικά ελλείμματα. Αυτό το ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητέ το πάνελ. Αυτό δείχνει ότι οι σταθεροποιητέ δεν λειτουργούν διότι οι δημοσιονομικοί κανόνες σημαίνει ότι οι χώρε που έχουν ύφεση έχουν μείωση εισοδημάτων και άρα εν τέλει πρέπει να κόψουν με τον ΑΒ τρόπο τα κοινωνικά επιδόματα. Αντί να υπάρχουν λοιπόν σταθερο θα στα, μειώνουν τα ήδη φυστάμενα πλαίσια. Τώρα, τι κινήσεις. Μπορεί να είναι κινήσεις από τις ε, φτωχότερες περιοχές, κινήσεις των πιο κινητών παραγόντων που μπορούν να μεριορίσουν την ανεργία με την έννοια ότι φεύγουν εργαζόμενοι αλλά μπορεί να έχεις προβλήματα διαθροτικής ανεργίας, που είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Φύγησε το να επιδείξω λίγο. Η ιδέα των ασυμμετρικών σοκ. Υπήρξαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν πολλά τέτοια συμμετρικά σοκ. Κάποια επηρέασαν τις, ανθρα... περιοχές με ορυχίες δεκαετία του 70 και του 80. Οι πρόσφατες περιλαμβάνονται εδώ πολλές. Η, κρίση στην Ασία με τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δημιού, επηρέασε πάρα πολύ τις ε, χώρες με εντατικοποίηση εργασίας όπως, αλλά λιγότερο Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα. Αυτά τα συμμετρικά σοκ επηρέασαν ισχυρά την ανταγωνιστικότητα των χωρών αυτών και τον 21ο αιώνα και νωρίτερα στη δεκαετία του 90. Η διεύρυνση είχε αρνητικές επιπτώσεις διότι έφερε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα με, χώρες με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ένωση που ανταγωνίζονταν ευθέω τις χώρες του Νότου. Ήταν πολύ καλό για την, ε, διεύρυνση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση η διεύρυνση, το γεγονός ωστόσο ότι ε, μπορούσαν να φύγουν επιχειρήσεις από τη μία χώρα σε και να εγκατασταθούν στην άλλη ήταν αρνητικό. Μεταξύ του 7 και του 12 η κρίση επηρέασε με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες χώρες. Επιπλέον δε... The monetary policy for countries with the current account deficit, which were most of the southern European countries, with either... Ε, θέλω να ανασφερθώ στο ότι σε μια νορμάλ κατάσταση η αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να γίνει με ε, υποτίμηση που δεν έγινε. Χώρες δηλαδή που είχαν ανταγωνιστικό πρόβλημα με χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία έχουν να αντιμετωπίσουν και μια ανατίμηση του ευρώ που ήταν ένα άλλο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των χωρών. Οι κεντρικοί σταθεροποιητές χρειάζονται διότι τα συμμετρικά σοκ υπάρχουν και μπορεί να είναι σκληρά προς τις χώρες. Τα κράτη-μέλη έχασαν πολλά εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης, ε, νομισματική πολιτική, ενώ οι περιορισμοί στην δημοσιονομική πολιτική σημαίνει ότι ε, χώρες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκυκλικές μακροοικονομικές πολιτικές, ενώ οι παράγοντες, ε, ε, οι κινήσεις των παραγόντων μέσα στην ενιαία ζώνη μπορούν να διευρύνουν τα, τα σοκ. Πρέπει να σκεφτείτε την περίπτωση διαθροτικών, διαθροτικής ανεργίας, ε, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμα, μεγαλύτερα, ακόμα πιο αρνητικές. Χρειάζονται λοιπόν κεντρικά αυτοματοποιημένοι σταθεροποιητέ, για να επιτρέψουν λίγο χώρο στους σταθεροποιητέ μέσα στου περιορισμού του ενίου νομίσματο και να αποφύγουν η οικονομική κρίση να οδηγήσει σε δημοσιονομική κρίση και χρηματοοικονομική κρίση, αποφεύγοντας και τα σοκ αυτά να οδηγήσουν σε μεγάλες περιόδους αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό έγινε στο επίπεδο του ΑΕΠ και της σύγκρισης με βάση τα στοιχεία της Eurostat από το 2001 και το 2007. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι χώρες με χαμηλότερα κατακεφαλήν εισοδήματα είχαν συγκλίνει με τις άλλες ε, χώρες της Ευρωζώνης τα τελευταία πέντε χρόνια και αυτό και το σενάριο των επομένων ετών έχει ένα Σαφέ σενάριο απόκληση των χωρών με τα χαμηλότερα εισοδήματα και αυτό είναι ο κίνδυνο τη μη ύπαρξη σταθεροποιητών και μη ύπαρξη συντονισμού των μακροοικονομικών πολιτικών που χρειάζεται η Ευρώπη. Θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε έτσι το πρώτο τμήμα της ακρόασής μας, δηλαδή γιατί χρειαζόμαστε αυτόματους σταθεροποιητές. Ε, γιατί χρειάζεται αυτό στην Ευρωζώνη και νομίζω ότι και οι τέσσερις ομιλητές ε, προέρχονται από background μακροοικονομικό και μας λένε ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος ε, της δημοσιονομικής προσαρμογής περιγράφει με ακρίβεια από τους τέσσερις ομιλητές. Έκανα τη διάγνωσή τους. Υπάρχουν ερωτήσεις Αλεχάνδρο Σέρκας και ποιος άλλος θα ήθελε το... Στίβεν Χιούς. Σαρές Άγια, η κυρία Παπαδοπούλου. Ωραία. Ε, ξεκινούμε με τον Αλεχάνδρο Σέρκας και, και ε, Σαρία Αγία και Ελιζαμπέτ Σρόντερ. Είστε ο συντονιστής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Μία, τον κύριο Φίσερ. Μάλιστα ο κύριο Όλια δεν ήθελα να την κάνω, αλλά και το έκανα δηλαδή, αλλά δεν μου απάντησε. Η ερώτηση είναι απλή κύριε Φίσερ. Ακούσατε, βάλατε ακουστικά, με ακούτε, με καταλαβαίνετε. Έλεγα, Φίσερ, ότι ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση που θα ήθελα να την κάνω στον κύριο Ριρέν και την έκανα αλλά δεν μου απάντησε. Μιλάμε γιατί παρότι μιλάμε συνεχώς για, αυτό, για ε, σταθεροποιητές, η Επιτροπή ουδέποτε το θέτει. Πώς συζητεί το θέμα αυτό στο κολέγιο. Εμείς λέμε αντί να συστήσουμε στα κράτη-μέλη να διαφυλάσσουν ως θησαυρό τους σταθεροποιητέ που έχουμε σε εθνικό επίπεδο, οι Βρυξέλλε από την άλλη μεριά δεν προσφέρουν στα κράτη που υφίστανται την κρίση καμία μορφή σταθεροποιητή, ενώ του συστήνει να καταστρέψουν και τους σταθεροποιητέ που έχουν σε εθνικό επίπεδο. Πώς το διαμορφώνει αυτό, κύριε Φίσερ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσάγια Σέντρικ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρουμε όλοι ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ε, και τα ε, επιδόματα ανεργίας ε, στα κράτη-μέλη χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους. Ρωτώ το εξής. Πώς θα γίνει αποδεκτό αυτό από πολιτικής πλευράς, διότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που εισφέρουν συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό πολύ περισσότερο από άλλες χώρες. Ε, τι, πώς πιστεύετε ότι θα τοποθετηθούν για αυτή τη μεταφορά πιστώσεων στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και ε, θεωρείτε ότι αυτό συνοβέλεται τρόπο τρόπος ώστε με κάποιον τρόπο να γίνει απόπειρα κάλυψης του χάσματος ανάμεσα στις βόρειες και τις νότιες χώρες της Ευρωζώνης. Ε, ευρύτατο αυτό που ρωτάτε. Αντιγόνη Παπαδοπούλου από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, είστε Κυπρία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ πλήρως τι σημαίνει αυτόματος σταθεροποιητής. Και ε, είμαι Κύπρια. Με το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι τράπεζες της Κύπρου, το Eurogroup επέβαλε μία λύση που ήταν κούρεμα ουσιαστικά επειδή δεν υπήρχαν αυτόματοι σταθεροποιητέ, επειδή δεν μπορούσε η Κύπρος που είναι μια μικρή χώρα στην Ευρωζώνη να εφαρμόσει δική της πολιτική για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Ανεργία, διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό, κοινωνικά προβλήματα και ειλικρινά δεν ρωτούμε, συμφωνώ με τον προβληματισμό του κυρίου Σέρκας, εκ των υστέρων ακούμε για τους αυτόματους σταθεροποιητές Αυτά όλα δεν τα σκέφτηκε το Eurogroup, δεν τα γνώριζε η Κομισιόν, δεν τα γνώριζε η Τρόικα. Γιατί αναγκαζόμαστε να καταστρέψουμε χώρες των Ευρωπαϊκών Νότων με τις άδικες πολιτικές λιτότητας της Τρόικας. Είδαμε προβληματικές πολιτικές στην Πορτογαλία και ύφεση. είδαμε παρόμοιες πολιτικές στην ισπανία στην ελλάδα σήμερα τη βιώνουμε στην κύπρο. αυτά όλα κατά την άποψή μου έπρεπε να υπάρχουν όταν οι χώρες έμπαιναν στην ευρωζώνη και απόλυσαν ουσιαστικά εθνική κυριαρχία και εργαλεία για να αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις. τώρα τι μπορεί να γίνει; στο διατάφτα πώς μπορούν αυτοί οι αυτόματοι σταθεροποιητές να διορθώσουν λάθη και τραγωδίες και κοινωνικές επιπτώσεις που ήδη τις βιώνουμε στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και ειδικά σήμερα στην Κύπρο. Χρειάζεται απάντηση για την κρίση ή μία λύση για το μέλλον. Ναι, νομίζω ότι αυτή η κρίση μας δίδαξε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους σταθεροποιητές είναι απαραίτητοι. Τους έχουμε παραγνωρίσει μέχρι τώρα. Θεωρήθηκε ότι οι νομισματικοί σταθεροποιητέ επαρκούν, αλλά μα αποδεικνύεται και με τα στοιχεία που φέρατε και του πίνακε ότι δεν επαρκεί βέβαια ε, να έχουμε μόνο οικονομικούς, νομισματικούς σταθεροποιητές. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν τέτοιοι σταθεροποιητές με, στο ιστορικό της χώρας πάντα μπορούν να λειτουργήσει επί παραδείγματι η φορολογία αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή φορολογική πολιτική δεν υπάρχει Πώς λοιπόν ε, θα βρούμε λύση χωρίς κοινή φορολογική πολιτική να εξασφαλίσουμε σταθεροποιητές κοινού. και επίσης χρειάζεται κοινή φορολογική πολιτική, είναι απαραίτητη και προϋπόθεση εκ των προκειμένου να, να υπάρξουν αυτοί οι σταθεροποιητές, να λειτουργήσουν ε, κοινοί σταθεροποιητές. Πρώτη ερώτηση και δεύτερη. Έχει προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ασφάλιση ενεργείας ή αντίστοιχες δυνατότητες. Ε, υπάρχουν όμως ε, μέτρα που θα μπορούσαν να μην πλήττουν τον ίδιο τον εργαζόμενο που είναι και η πιο αδύναμη ομάδα αλλά παραδείγματι μέτρα στα οποία θα μπορούσε με βάση εισοδηματική, με κριτήρια εισοδηματικά οι άλλες δυνατότητες να αναπτυχθούν σταθεροποιητές. Η Πρόεδρος. Έχετε δεχτεί μια απευθεία ερώτηση και θα πρέπει να απαντήσετε ασφαλώ και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι, αλλά πρέπει να περάσουμε και στην ουσία του ζητήματο, που θα είναι η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση που έχει διατυπώσει η Επιτροπή μα. Α ακούσουμε λοιπόν τον κύριο, τον κύριο Γκέορκ Φίσερ πρώτα και μετά οι υπόλοιποι. Λυπούμε, αλλά θα πρέπει να πω ότι εγώ δεν είμαι επίτροπος. Δεν ανήκω στο συλλογικό όργανο που ονομάζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του δεν τελώ εν γνώση των συζητήσεών τους. Ε, τίθεται πάντως το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το blueprint αυτό, με, την με το προσχέδιο, όχι όμως με τη μορφή πρότασης, δεν έχει προτείνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη. Το Συμβούλιο φαίνεται να σκοπεύει στο δεύτερο εξάμεινο να επανέλθει θα δούμε τι ε, τοποθέτηση θα προκύψει και πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως εμείς έχουμε θεσπίσει μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης για την Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Οικονομικών Νομισματικών Θεμάτων ε, μια ομάδα εργασίας η οποία έχει παραγάγει ε, τοποθετήσεις και εκθέσεις οι οποίες πιστεύω αποτελούν και τη βάση ε, τον όσο θα σας παρουσιάσουν αργότερα σήμερα οι Γερμανοί στην Αλφή. Δεν είναι δημοσιευμένα επισήμως αυτά, ωστόσο σε λίγο καιρό θα, θα τα δείτε στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης για την Απασχόληση. Υπάρχει δουλειά ακόμα που γίνεται, αλλά συγκεκριμένη πρόταση ακόμα δεν έχει κατευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό μπορώ να πω όμως ότι το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επεξεργάζεται το θέμα αυτό. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να δώσω σε πρώτη φάση. Τα υπόλοιπα στο δεύτερο κομμάτι της συζητήσεως. Ο κύριος λοιπόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα για τις δύο ερωτήσεις οι οποίες έχουν ε, κέριο χαρακτήρα, εάν είναι απαραίτητη δηλαδή η ύπαρξη σταθεροποιητών και αν ισοδυναμεί με τις μεταφορές κονδυλίων. Πρώτη ερώτηση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς την επιχειρηματολογία που θα προβάλλουμε για την ε, ασφάλιση ενέργειας, για τι αυστηρά οικονομικού όρους και προοπτικές, εάν ρωτήσει κανείς πώς είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν τα ασυμμετρικά αυτά πλήγματα για τα οποία συζητούμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ποσοτικά ο πρώτος διάβλος ε, κατανομής του, του κινδύνου είναι οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Μέσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορά μεταξύ Νεβάδας και Τέξτας και Τέξας δεν αντιμετωπίζεται με οικονομικές μεταφορές κονδυλίων από το κράτος, αλλά με την τραπεζική ένωση που υπάρχει και την ε, διαπολιτιακή μεταξύ δηλαδή των πολιτιών κυριότητα σε ε, περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή η Νεβάδα έχει ακίνητα στο Τέξας και, και Τούμπαλιν. Παράδειγμα. Όταν χάσει παραδείγματι ένα δολάριο η μία πολιτεία σε σχέση με την άλλη, το 46%, τα 46 cents θα τα καλύψει η χρηματοπιστωτική αγορά. Τα 25 θα τα καλύψει ο κρατικό προπολογισμό. Ο ομοσπονδιακό προπολογισμό. Και πέραν αυτού θα αρχίσουν να νοικιάζουν, να δανείζονται συγγνώμη, τα νοικοκυριά. Μοιράζονται και αυτά δηλαδή κάπως τον κίνδυνο. Ασφαλώς λοιπόν χρειάζεται το πρώτο, αναμφίβολα χρειάζεται το πρώτο, τραπεζική ένωση και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μετά όταν αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα σταθεροποιητικά, τότε ναι, αλλά στη δεύτερη φάση, και αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη για να είμαστε σαφείς, αυτό όμως είναι μόνο μία καθαρά οικονομική ανάλυση που σας εκθέτω. Μετά έρχεται η πολιτική ανάλυση. Και αυτή λέει ότι η Τραπεζική Ένωση έχει χαρακτήρα τεχνοκρατικό. Δεν είναι αντιληπτή για τον πολίτη καθαρά όπως ένα επίδομα ανεργίας. Και άρα έρχεται να δοθεί μια άλλη απάντηση πολιτική στην ερώτησή σας. Πάντως, οι μηχανισμοί αυτοί δεν χρειάζεται να είναι μακροπρόθεσμα μηχανισμοί μεταφοράς κονδυλίων. Δεν χρειάζεται. Μπορεί δηλαδή να σχεδιαστούν έτσι ώστε οι χώρε και να μοιράζονται του κινδύνου μένα, αλλά μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα 20-30 ετών να είναι μηδενικέ οι μεταφορέ. Πάλι πολιτική επιλογή. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ να συμπληρώσω κάποια πράγματα σε σχέση που αυτά που μόλις ακούσαμε, πρέπει να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα ε, στις κυκλικές ε, μεταφορές ε, πιστώσεων και τις διαρθρωτικές. Οι πρώτες χρησιμοποιούνται για την σταθεροποίηση των κυκλικών εξελίξεων της πραγματικής οικονομίας και δεν μπορούν να διορθώσουν μακροπρόθεσμες ανισορροπίες. Εάν αυτό χρησιμοποιηθεί ως αυτόματος σταθεροποιητής, γιατί όλοι αυτό έχουμε κατά νου, κατά τη διαστολή με ένα μόνιμο ε, σύστημα μεταφοράς πιστώσεων, δεν πρόκειται να διορθώσει την ανισορροπία στην Ευρωζώνη, ούτε και να λύσει το πρόβλημα που μας οδήγησε στην χρηματοοικονομική κρίση. Θα το είχε ελαφρύνει, θα το είχε μετριάσει το πρόβλημα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα με πάγιο τρόπο δεν θα είχε διορθώσει τι ανισορροπίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφή πρέπει να είναι η διάκριση ανάμεσα στις, ε, στην κυκλική αστάθεια και τη διαρθρωτικού χαρακτήρα αστάθεια και άρα ε, διαφορά ανάμεσα στις μεταφορές ε, πιστώσεων. Φυσικά αυτό όταν δεν υπάρχουν σοβαρέ αποκλήσει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θέλετε κι εσεί να προσθέσετε κάτι, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Καλντέρα Καμπράλ, θα ήθελα να προσθέσω κάτι στη συζήτηση. Η Τραπεζική Ένωση θα είναι πολύ σημαντικότερη για κοινωνικά ζητήματα από ότι μερικοί μη οικονομολόγοι που και που το θεωρούν. Το βασικό θέμα είναι το θέμα των καθαρών πληρωτών, των καθαρών δικαιούχων και οι μεταφορές κονδυλίων από βορρά προς νότο. Θα πρέπει να σας πω ότι τα προσωρινά μέτρα δεν χρειάζεται μόνιμα. Αν δείτε, όπως αναφέρθηκα προηγουμένως, το επίπεδο ανεργίας στα διάφορα κράτη της Ένωσης, το παράδειγμα της Πορτογαλίας, για παράδειγμα, είναι καλό. γιατί τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και αργότερα ήταν κάτω από το μέσο όρο. Ε, λοιπόν από το σύστημα. Δεν θα υποφελεί το μάλλον από το νέο σύστημα. Τώρα θα υποφεληθεί. Άλλες χώρες της Ένωσης που είχαν υψηλή ανεργία στο παρελθόν ή κάποιες περιφέρειες που επηρεαστούν στο μέλλον μπορεί να κερδίσουν. Άρα είναι ένας καταμερισμός κινδύνου που θα βοηθήσει κάποιες χώρες ή κάποιες περιφέρειες τώρα όπως βοήθησε κάποιες χώρες ή κάποιες περιφέρειες στο παρελθόν. Να τονίσω επίσης ότι υπάρχουν μεταβιβάσεις στο εσωτερικό της Ένωσης. Στη γεωργία, στα διαφθορτικά ταμεία, στις μεταφορές στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές το μεγάλο πρόβλημα που όλοι εντοπίζουμε στην Ευρώπη σήμερα είναι η ανεργία. Οι μεταφορές λοιπόν, οι μεταβιβάσεις σε περιφέρειες με υψηλή ανεργία είναι λογικές στο πλαίσιο της ευρύτερης επισκόπησης της Ευρώπης. Ιδίως αν είναι βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα για χώρες με μεγάλη ανεργία τώρα. Είναι λογικό να χρησιμοποιήσεις ε, αυτές τις διαδικασίες τώρα και καθιστά εύλογη τη μεταφορά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολία, δυσκολίες. Δυσκολίες που δημιουργούνται από την έλλειψη εργαλείων που προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Επίσης επιδεινώνονται από την έλλειψη συντονισμού δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών που είναι όλες σε φάση λυσότητας, ενώ άλλες δεν είναι. Είναι λάθος δηλαδή να πιστεύουμε ότι τέτοιες μεταβιβάσεις δεν είναι εφικτές ενώ είναι. Οι σταθεροποιητές μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία αλλά προφανώς με ε, Δεύτερη ερώτηση. Τι κάνουμε και πώς εμείς διαπραγματευόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους. Ένα θέμα επικουρικό, αλλά πρέπει πρώτα να ε, δούμε τι, ποια δράση χρειάζεται. Κύριε Φίσερ, προσέξτε, καταρχάς αυτό δεν είναι λύση για τα πάντα. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές. Αν δεν υπάρξει τραπεζική ένωση, μάλλον θα μας ε, ε, βοηθήσει λίγο. Και αυτό, αυτή την προσέγγιση ακολουθεί το blueprint. Ε, η Κομισιόν στο blueprint περιλαμβάνει μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο φάσμα μέτρων που μπορούν να βοηθήσουν. Κατά βάση υπάρχουν δύο εναλλακτικέ και στη βιβλιογραφία και στην πράξη. Ένα, μακροοικονομικό εργαλείο σταθεροποίησης, αυτό που ανέφερε εσύ. Έχει το πλεονέκτημα ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση και το μειονέκτημα ότι θα είναι δύσκολο να εξηγηθεί σε κάποιον πέραν κάποιων μακροοικονομολόγων. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι λειτουργεί με έναν δίκτυ παραγωγή, με βάση το δίκτυο παραγωγή, που δεν είναι σταθερό, αλλά τέλο πάντων μπορεί να το λύσουμε. Ο δεύτερο υποσυζήτηση μηχανισμό σχετίζεται με την ενεργεία, με τα επιδόματα ενεργεία. Συμφωνώ ότι υπάρχει ένα στοιχείο οικονομική ορθολογική, διότι η πάρα εξαρτάται πάρα πολύ από οικονομικού κύκλου. Υπάρχει ωστόσο και ένα στοιχείο πολιτική και κοινωνική πολιτική. Αυτό είναι δεδομένο. Αν οι αποφάσεις ε, ληφθούν μπορεί να παρακολουθήσουν και, τις δύο, και τους δύο προσανατολισμούς. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι και στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει ένα αντίστοιχο σύστημα που έχουν με αντίστοιχη μίξη πολιτικών και οικονομικών λόγων. Συνεχίζοντας, το σύστημα που περιγράφεται λίγο στην βιβλιογραφία είναι ένα σύστημα που περιγράφεται και στο blueprint και που πρέπει να είναι ανοιχτό, εύκολο, προσωρινό και να προωθεί την αλλαγή. Διότι προφανώς μπορούμε να φτιάξουμε σύνθετα συστήματα, αλλά έχουμε 28 κράτη με δικά τους εθνικά συστήματα επιδοτήσεων ανεργίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να ξεκινήσουμε εξ αρχής. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ταιριάζει στη δομή της Ένωσης. Το σύστημα λοιπόν της Ένωσης θα πρέπει να είναι ελαφρύ, προσωρινό, διάφανο και να προωθεί την, αλλαγή, την Προσωπικά, και το λέω σαφώς, η άποψή μου είναι ότι ένα σύστημα που στηρίζεται σε επιδόματα ενεργείες θα έπρεπε να καλύπτει αυτές τις τέσσερις προϋποθέσεις. Μπορώ να... Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, θα σας πάρω πολύ χρόνο. Να σταθώ ωστόσο σε αυτό το σημείο της διαφάνειας η ανεργία είναι κάτι που καταλαβαίνει ο κόσμος. Βλέπουν τον άνεργο στο δρόμο, βλέπουν τους αριθμούς των ανέργων, ξέρουν ότι ο κόσμος γίνεται ανέργος. Κάποια μορφή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ε, ΟΝΕ θα είναι κατανοητό, θα είναι κατανοητή. Για το ερώτημα τώρα από τις σκανδιναβικές χώρες. Αν δούμε τα νούμερα, ιστορικά, θα υπήρχε μία περίοδος όπου χώρες όπως η Γερμανία ή η Σουηδία, αν ήταν τότε μέλος της ΟΝΕ, θα είχαν επωφεληθεί από ένα τέτοιο σύστημα. Προφανώς είναι σαφές ότι ε, οι χώρες που θα κερδίσουν είναι χώρες με τη μεγάλη ανεργία, αλλά στην ιστορικά έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες και στη Γερμανία είχε υψηλή ανεργία. Μην ξεχνάτε ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε την ποιότητα ενός συστήματος μόνο από το τι βλέπουμε σήμερα. Αυτό θέλω να το τονίσω. Αν δείτε το σύστημα ανεργίας ε, στη Γερμανία, στην Αυστρία, θα δείτε ότι σε συγκεκριμένους ε, χρόνους, συγκεκριμένες περιφέρειες της Αυστρίας ή της Γερμανίας κέρδισαν από το σύστημα αυτό, διότι το οικονομικό κλίμα με, αλλάζει και υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτό έτσι πάντα. Κάτι ακόμα και τελειώνω. Η πρόθεση της αλλαγής. Και τώρα ένα πλεονέκτημα των ε, συστημάτων αυτών είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις, γι' αυτό λέω μπορεί, για να δουν και πώς τα συστήματα επιδομάτων ενεργείας και τα συστήματα ενεργής παρέμβασης στην αγορά εργασίας λειτουργούν στα κράτη. Αυτό μπορεί να το δει κάποιος ή να μην το δει για καθαρά οικονομικούς λόγους, αλλά μάλλον θα γίνουν διότι εν τέλει θα θέλαμε να έχουμε ένα σύστημα που να ωφελεί αυτούς που το χρειάζονται. Αν έχουμε διαφορές στο σύστημα κάλυψης των ανέργων από 30% έως 85% στις χώρες ΩΝΕ, θα τεθεί το ερώτημα, αρκεί το 30% για να πετύχεις ε, την οικονομική κοινωνική λειτουργία που θέλει. Θα σταματήσω εδώ ωστόσο. Um, Yes, so, so on the, uh, on the question of, of uh, how... Για το πώς, το θέμα του πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπατε. Δύο είναι οι στόχοι. Ο ένας είναι αμυγός οικονομικός και ο άλλος είναι κοινωνικό-πολιτικός. Ο οικονομικός στόχος από μόνος του δεν επαρκεί, δεν είναι επαρκές κίνητρο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο επιμερισμός κινδύνων σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές αγορές, μόνο και μόνο από άποψη οικονομικών μεγεθών. Από εκεί ξεκινάμε, αλλά δεν επαρκεί. Υπάρχει αυτή η πολύ ισχυρή κοινωνικοπολιτική διάσταση και όλοι θα συμφωνήσετε, νομίζω. Κατά τον σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος, το κλειδί είναι η απλότητα. Γι' αυτό μ' αρέσει αυτή η ιδέα της ασφάλισης και ο Πιέρ Μουσκοβίτσι γι' αυτό το λόγο μεταξύ άλλων πρότεινε ένα τέτοιο πρότυπο ε, στα πλαίσια ενός προϋπολογισμού για την Ένωση αυτό το σύστημα ασφάλισης. Το λέω αυτό για να καταλάβουν όλοι περί τίνος πρόκειται. και ε, να επανέλθω σε αυτό που με ρωτήσατε για το χάσμα ανάμεσα στις βόρειες και τις νότιες χώρες. Δύο είναι τα ζητήματα. Είναι μηχανισμός ε, μεταφοράς ε, πιστώσεων πρώτον και δεύτερον. Ποια είναι τα κίνητρα για να γίνουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές είναι οι βασικές ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε. Είναι ένα σύστημα μεταφοράς Εξαρτάται από το σχεδιασμό θα σας απαντήσω. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικά ποσοστά ανεργίας. Μπορείτε να πάρετε το μέσο όρο. Ε, είναι προφανές ότι στην Ισπανία είναι πολύ υψηλότερος ο μέσο όρος ακόμη και στο, την ίδια στιγμή του ε, οικονομικού κύκλου. Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόκληση από το μέσο όρο. Δηλαδή η ροή των πιστώσεων θα είναι συνάρτηση του μέσου όρου του ποσοστού ανεργίας της χώρας. Πώς γίνεται αυτό. Για να παραμείνουμε απλοί, γιατί αυτό είναι το κλειδί, οι δικαιούχοι των επιδομάτων δεν πρέπει να ασχοληθούν με το από πού θα λαμβάνουν το επίδομα, θα πρέπει να ξέρουν ότι ε, το επίδομά τους προέρχεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και κάθε ή κάθε μία άνεργος ε, θα λαμβάνει αυτό το επίδομα μπορείτε να ξεκινήσετε δοκιμαστικά με τους νέους. Αλλά πώς χρηματοδοτείται ένα τέτοιο σύστημα όταν το επίπεδο της χρηματοδότησης εξαρτάται από το μέσο όρο του ποσοστού ανεργίας της κάθε χώρας. Εάν λοιπόν πλησιάζουν ε, το μέσο όρο τα περισσότερα κράτη-μέλη, δεν θα υπάρχουν ε, καθαρές ροές, δηλαδή θα εκταμιεύουν και θα εισπράττουν περίπου τα ίδια ποσά τα κράτη-μέλη. Δείτε όμως ένα στιγμιότυπο του 2005, παραδείγματος χάρη. θα, ήταν πολύ κάτω από το μέσο όρο, το αντίθετο συμβαίνει στην ε, Γερμανία, οπότε υπάρχει καθαρή ροή πιστώσεων από την Ισπανία προς τη Γερμανία με αυτό το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σήμερα ε, θα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Μην ξεχνάμε ότι ε, από το 1,5 πέρασε η Ισπανία στο 3% του ΑΕΠ για τα επιδόμετα ε, ε, ε, ανεργίας. Δηλαδή, μια μισή μονάδα. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Ίσως να καλυφθεί κατά το ίμιση. Ε, και να καλύψετε κάτι ανάμεσα στο μισό, στη μισή και τη μία ποσοστία μονάδα. Η πολλαπλασιαστές της κρίση τώρα, δηλαδή η επίπτωση της κρίσης επί της ανάπτυξης, ε, μας οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα για τη σταθεροποίηση, όχι ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε ένα τέτοιο σύστημα, οι ροές ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ισπανία θα είναι μηδενικέ σχεδόν. Αυτό πρέπει να το συμπολογίσουμε όταν σχεδιάζουμε το σύστημα. Για τα κίνητρα τώρα. Επίσης είναι ένα θέμα κλειδί, διότι το αντεπιχείρημα κατά ενός συστήματος επιμερισμού κινδύνου είναι ακριβώς ότι θα μειωθούν τα κίνητρα ε, για να διεξαγάγουν τις σωστές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη, οι οποίες ε, θα οδηγήσουν σε μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. Ε, κατά τη γνώμη μου, ποια είναι η απάντηση. Φυσικά, μπορούμε να πούμε, όπως σας περιέγραψα το, τη μεταφορά πιστώσεων, ε, το κυκλικό κομμάτι συνεπάγεται ότι παραμένουν τα κίνητρα για τα κράτη-μέλη για να μειωθεί η διαρθρωτικού τύπου ανεργία, διότι δεν καλύπτεται από αυτό το σύστημα. Οπότε έχουν κάτι συμφέρον να το κάνουν. Όμως αν παραμένει, πάγια σε υψηλό επίπεδο, αν αποκλίνετε πολύ, θα πληρώσετε υπερβολικά πολλά χρήματα για να καλύψετε το κενό. Οπότε και αυτό είναι ένα κίνητρο για να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία. Δεύτερον, μπορείτε να επιλέξετε να αρχίσετε με ένα είδος ανεργίας που είναι μάλλον, συνδέεται μάλλον με την έλλειψη τύχης, ε, πολύ κακό μακροοικονομικό φαινόμενο. Καλό σημείο κίνησης θα ήταν οι νέοι άνεργοι και ίσως να υπάρχει μια περιορισμένη χρονική περίοδος για το σύστημα ασφάλισης. Αυτό έχει τα μειονεκτήματά του, αλλά τουλάχιστον κρατάει ζωντανά τα κίνητρα. Για το ποσοστό αναπλήρωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει ένα βασικό επίπεδο και τα κράτη-μέλη που θέλουν να είναι πιο γενναιόδωρα έχουν την επιλογή, μπορούν να υπερβούν αυτό το ποσοστό. Θα έχετε ένα νέο περιθώριο. Αν ένα κράτο ε, επιλέξει να είναι πιο γενναιόδωρο, ε, λοιπόν θα πληρώσει από την τσέπη του τα ε, επιπρόσθετα ευρώ. Έχουμε ένα αρχικό επίπεδο αποζημίωσης και ας πάρουμε μία 9 μηνή ή 12 περίοδο αποζημίωσης. Νομίζω ότι αυτά επαρκούν τόσο ώστε να παραμείνουν εν ζωή τα οικονομικά κίνητρα που θα έχουμε θεσπίσει κάτω το του προγράμματος. Ευχαριστούμε λέει αλλά έσβησε το μικρόφωνο της. ο κύριος Φίσε. Ε, ουσιαστικά Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα για αυτό που μας είπε ο κύριος Φίσερ. Δύο είναι οι ιδέες, δύο είναι οι δυνατότητες ε, για αυτούς τους αυτόματος σταθεροποιητές. Ε, είτε να έχουμε μεταφορά ε, πιστώσεων και να το συνδέσουμε με τις αποκλήσεις ανάμεσα στην πραγματική η οικονομική κατάσταση όταν ε, δουλεύει με πλήρη ρυθμό, ε, με πλήρες τροφές ε, και την πραγματική οικονομική κατάσταση. Δηλαδή είναι όταν έχετε αρνητικό χάσμα ως προς το output, ως προς τα αποτελέσματα σε σχέση με το πραγματικό δυναμικό της χώρας, τότε θα λαμβάνει επιστώσεις από μια χώρα που έχει θετικό τέτοιο δίκτυο, έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το πραγματικό δυναμικό της. Εάν αυτό το σύστημα μεταφοράς βασίζεται στις επιδόσεις των κρατών μελών, θα μας οδηγήσει σε ένα τέτοιο σύστημα. Αν δούμε τώρα τη διαφάνεια, βλέπουμε την απόκληση αποτελεσμάτων, output gap για τη Γερμανία, αν δείτε στις διάφορες χρονικές στιγμές όπου γίνεται η αποτίμηση, βλέπετε φοβερές αλλαγές και διακυμάνσεις σε αυτό το χάσμα. Ίσως δεν μπορείτε να το διαπιστώσετε, αλλά υπάρχουν διαφορετικές χρειές πράσινου που δείχνουν τα αποτελέσματα που έχει δημοσιεύσει ο ΩΣΑ, παραδείγματο χάρη, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπίπτουν τα νούμερα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν μαζικέ αποκλήσει ω προ τι αξιολογήσει του χάσματο αποτελεσμάτων, ανάλογα με το αν έγινε η αποτίμηση νωρίτερα στο χρόνο, εάν θα και αυτό ότι αν χρησιμοποιηθεί αυτό το μέγεθος ως βάση για τον υπολογισμό, ενδέχεται να υπάρξει πολιτική παρέμβαση σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Αν δούμε το σύστημα ασφάλισης για την Ισπανία, κοιτάξτε αυτή τη διαφάνεια, βλέπουμε επίσης πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις ε, σύν το χρόνο κατά την αποτίμηση ε, της διαφοράς αποτελεσμάτων. Δεν είναι αρκετά αξιόπιστο μέγεθος για να χρησιμοποιηθεί ως βάση, διότι με το χρόνο ή μάλλον να το πω έτσι, ή πρέπει να περιμένετε για ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα, οπότε όμως θα έχουμε ξεφύγει από τον οικονομικό κύκλο και δεν θα είναι δυνατή η μεταφορά των πιστώσεων, ή θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης, όπως είπε ο κ. Φιλίπ ε, Ντυπού, θα μπορούσαμε να βασίσουμε το σύστημα ε, στις αποκλήσεις από έναν μέσο όρο ανεργίας. Οι κυκλικές διακυμάνσεις του ποσοστού ανεργίας πρέπει να διαφοροποιηθούν από τις ε, διακυμάνσεις, τις διαρθρωτικές ανεργίες. Όμως η βραχυπρόθεσμη ανεργία είναι αυτή που είναι η προκυκλική, η μακροχρόνια. Πάνω από τους 12 μήνες είναι διαρθρωτικού τύπου ανεργία. Αν όμως επικεντρωθούμε στη βραχυπρόθεσμη ανεργία μέχρι τους 12 μήνες, τότε πάνω κάτω γίνεται αυτόματα αυτή η διάκριση ανάμεσα στην στις κυκλικού χαρακτήρα και διαρθρωτικού χαρακτήρα αποκλήσεις. Προτείνουμε το εξής λοιπόν. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης που δίνει ένα βασικό επίδομα ανεργία σε όλες τις χώρες και αν οι εθνικές κυβερνήσεις αποφασίσουν ότι επιθυμούν να έχουν ένα βελτιστοποιημένο ε, σύστημα ασφάλισης υπέρ αυτού του ευρωπαϊκού, πολύ βασικού ομολογουμένου επίπεδου αποζημίωση, είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής. Εάν λοιπόν οι εθνικές κυβερ... κυβερνήσεις αποφασίσουν ότι θέλουν για... Ε, να είναι πιο γενναιόδορες μπορούν να δώσουν μια προσάυξηση. Γι' αυτό έχω χρωματίσει με πράσινο αυτή τη ζώνη. Βλέπουμε το επίδομα ανεργία στο ευρωπαϊκό που, που είναι ευέλικτο, αλλά το συγκεκριμένο παράδειγμα καλύπτει 12 μήνη περίοδο ανεργίας. Οτιδήποτε υπερβαίνει αυτούς τους 12 μήνες πρέπει να καλυφθεί αυτόματα από το εθνικό σύστημα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια ως προς τα επιδόματα είναι το 50% του τελευταίου μισθού και αν η κυβέρνηση ενός κράτους θέλει να ε, δώσει μια προσάυξηση και να έχει υψηλότερο επίδομα ανεργίας, μπορεί, έχει τη δυνατότητα να το πράξει. Είναι εντελώς ευέλικτο αυτό το σύστημα. Μπορείτε να αυξομειώνετε την ευρωπαϊκή συνιστόσα του επιδόματος ενεργείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καλύψετε όλες τις περιπτώσεις. Οτιδήποτε ε, εκπίπτει της ευρωπαϊκής διάστασης καλύπτεται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Είναι μάλλον προφανές ότι ε, χρειάζεται αυτόματο σταθεροποιητή, διότι όπως και στο εθνικό επίπεδο, πάντοτε έχετε μεταφορές πιστώσεων από αυτού που έχουν δουλειά προς αυτούς που δεν έχουν ακόμη και σε εθνικό επίπεδο. Αυτοί συνεισφέρουν όσοι έχουν μια θέση απασχόληση και οι υπόλοιποι είναι δικαιούχοι και λαμβάνουν το επίδομα ανεργία ακριβώ επειδή δεν έχουν. Υπάρχει μεταφορά ούτω ή άλλω. Δεν υπάρχει όμω πολιτική παρέμβαση. Δεν χρειάζεται μια επιτροπή που θα αποφασίσει πότε θα γίνουν οι μεταφορέ ανάμεσα στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Υπάρχουν και άλλα πλέον εκτήματα. Είναι σχετικά απλό ε, να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα εθνικά συστήματα για, να, ε, για τη συλλογή των εισφορών και την καταβολή των ε, επιδομάτων. Δεν χρειάζεται μία υπερεθνική αρχή που θα αποφασίζει ποιος είναι άνεργος, ποιος είναι επιλέξιμος και ποιος όχι. Οι εθνικοί οργανισμοί θα το αποφασίζουν. Επίσης πρέπει να είναι η μεταφορά μάλλον κυκλικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί να έχει πάγιο χαρακτήρα. Σε κάποιες χώρες, και αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε, θα ε, ε, λαμβάνουν ε, για μεγάλη χρονική περίοδο εισφορές. Βλέπουμε τις αποκλήσεις από το μέσο όρο του ποσοστού ανεργίας της Ευρωζώνης εδώ για κάποιες χώρες. παράδειγμα χάρη, ο κύριο Φίσερ αυτό μας έλεγε. Ακόμη και η Γερμανία θα ήταν δικαιούχος ε, για ένα τέτοιο επίδομα, διότι σε κάποια στιγμή το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία ξεπερνούσε το μέσο όρο ε, της ανεργίας στην Ευρωζώνη. Ποιο είναι το πρόβλημα. Η περίπτωση της Ισπανίας. Δείτε εδώ, ήταν υψηλότερο το ποσοστό ανεργίας ε, για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπου ήταν στην ε, νομισματική ένωση. Παρότι ήταν σχετικά καλά η οικονομική κατάστασή της, ε, είχε υπερθερμανθεί η οικονομία και υπήρχαν και οι μεταφορές από ένα τέτοιο σύστημα θα είχαν ως αποτέλεσμα αφαίρεση της αγοραστικής δύναμης της Ισπανίας και μεταφορά αυτής σε άλλες χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό θέλουμε να τα αποφύγουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουμε τα οικονομικά μεγέθη. Είναι λίγο δύσκολο να κρίνουμε εκ των προτέρων ε, είτε το κόστος είτε το κατά πόσο θα λειτουργήσει αυτός ο σταθεροποιητικός παράγοντας ε, ή Ποιο, ποια ποσά, ποιες εισφορές χρειαζόμαστε, θα είναι υπέρ του 1,5% του ακαθάριστου μισθού. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό, ξαναλέω, λειτουργεί συμπληρωματικά με τα εθνικά συστήματα. Ε, ε, δηλαδή το ίδιο ποσό θα πηγαίνει στον ε, κορβανά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα λειτουργεί, ξαναλέω, συμπληρωματικά σε σχέση με τα εθνικά συστήματα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να σας δώσω λεπτομέρειες, όμως υπάρχουν άρθρα και τα αναφέρω σε σχέση με τους σταθεροποιητές και να προσθέσω και κάτι τελευταίο γιατί αναφέρθηκε προηγουμένως. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα είχαμε αναχαιτήσει ή σταματήσει την κρίση, αλλά μετριάζουμε τον αντίκτυπό της. Υπολογίσαμε ότι το η σταθεροποίηση στην Ισπανία θα ανερχόταν στο 20% αν είχαμε το 2008 και 2009 ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα και ε, θα κειμενόταν στο 20% η σταθεροποίηση δηλαδή θα είχαμε μειώσει τη μείωση του ΑΕΠ κατά 20% εάν το 2008 μέχρι το 2010 είχαμε ένα τέτοιο σύστημα και για την Ιρλανδία και την Ελλάδα ε, αυτό, αυτή η σταθεροποίηση θα κειμενόταν περίπου περίπου στο 10% για την ίδια χρονική περίοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Μπορείτε να βάλετε τη δική μου παρουσίαση PowerPoint, σας παρακαλώ. Δεν μελέτησα το, με τόσο εντελεχή τρόπο τον αντίκτυπο της κρίσης, αλλά μπορώ να σας δώσω κάποιες ιδέες οι οποίες που είναι μάλλον ε, χαμηλότερο προφίλ. Μιλήσαμε για την δυνατότητα ίδρυσης ενός ασφαλιστικού ταμείου. Όπως αυτό που προτάθηκε νωρίτερα μάλλον. Συμφωνώ, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά. Η εναλλακτική λύση θα ήταν σε περίπτωση υπέρβασης του κατοφλίου, αντί να έχουμε μαζικές πιστώσεις, η αναλλακτική, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι καλύτερη. Κάποιες χώρες θα λάμβαναν αυτές τις πιστώσεις και το βασικό ζήτημα θα ήταν πώς μετράτε η ανεργία και κατά πόσο ξεπερνάτε ο μέσος όρος της ανεργίας από κάποια κράτη-μέλη και ε, κατά πόσο το ποσοστό ανεργίας και αυξομοιώσεις του συσχετίζεται με το output gap, τη διαφορά ανάμεσα στις οικονομικές επιδόσεις ε, των κρατών. Όταν μιλάμε για ποσοστό 12% ανεργίας και διαφορές σε δύο τριών ποσοστίων μονάδων σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, θα ήταν καλή εναλλακτική λύση ένα τέτοιο σύστημα. Όμως, θα έπρεπε να υπάρχουν όλα αυτά στην αρχή της αιρεσιμότητας, να βρούμε τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα και εάν λαμβάνουν στήριξη κάποια κράτη-μέλη λόγω υψηλής ανεργίας, τότε θα οπίσουμε το θέμα της μεταφοράς των πιστώσεων μέσα από τα επιδόματα ανεργία, δηλαδή να διαπιστώσουμε αν αυτό σχετίζεται με την αρχιτεκτονική του συστήματος κοινωνική προστασία. Μία αιρεσιμότητα σε εθνικό επίπεδο πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογιστεί κατά το σχεδιασμό του συστήματος, Αλλιώ θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει δεκτό από πολιτική σκοπιά το σύστημα. Αναθεώρηση βλέπουμε της νομοθεσίας. Ε, θα μπορούσε να τεθεί και αυτό το ζήτημα εάν Μιλάμε για τις μεταφορές πιστώσεων για την απευθεία στήριξη των ανέργων. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι ομοιόμορφο το σύστημα, όμως, όπως ακούσαμε, αν θέλουν κάποιες χώρες να είναι πιο γενναιόδορες, δεν πρέπει να καταβάλουν το τίμημα όλα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν επιλέξει να έχουν τόσο γενναιόδορα συστήματα κοινωνικής ε, ασφάλισης. Μια άλλη ιδέα θα ήταν, αλλά είναι λίγο διαφορετικό αυτό το σύστημα, να έχουμε ένα επίδομα ανεργίας σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα λειτουργούσε ως βασικός οικονομικός σταθεροποιητής ε, και να έχουμε μεγαλύτερη παρέμβαση σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής για τις περιοχές που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Άρα θα πρέπει να έχουν κονδύλια για επενδύσεις, για απευθείας ε, για απασχόληση κτλ. Ε, όλα αυτά υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν και αυτός είναι ένας ε, πιο ελαφρύς τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση κάπως. Έτσι λοιπόν, στα διαφορετικά ταμεία θα πρέπει να ενσωματωθεί ένα ταμείο απασχόλησης, κάτι που θα ενεργοποιείται από ένα επίπεδο ανεργίας, δύο-τρεις μονάδες, σε παραδείγματι, πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, και θα καλύπτει για δύο, τρία ή πέντε χρόνια με προσωρινά μέτρα στην αριστερή παρέμβαση, παραδείγματι υποστήριξη για επενδύσει, υποστήριξη στην κατάρτιση, πέραν των διαρθρωτικών ταμείων που υπάρχουν. Και ένα άλλο τρόπο το κοιτάξουμε αυτό. Με τους στόχους και τα προγράμματα των ταμείων που ήδη υπάρχουν, θα ήταν η απασχόληση να οριστεί ως προϋπόθεση για την ενίσχυση της, ή την επιτάχυνση της πρόσβασης στα κονδύλια ή την εμπροστοβαρή αξιοποίηση των κονδυλίων. Και αυτό ήταν ένας πολύ ε, απλός τρόπος για την αξιοποίηση σταθεροποιητών, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ γρήγορα. Επί παραδείγματι, περιοχές που έχουν σημαντική ενεργεία μπορούν να μετατρέπονται σε περιφέρειες στόχου 1, εάν είναι ως προς το εισόδημα κοντά στο μέσο όρο. Εάν έχουν και χαμηλότερο από το μέσο όρο εισόδημα και υψηλή ανεργία, τότε θα πρέπει να τους δίδεται από τα κονδύλια αυτά ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως η εναλλακτική που προτείνουμε είναι η επιπλέον αξιοποίηση, η μεγέθυνση των μέσων που υπάρχουν ήδη ή η εστίαση τους περισσότερο στις περιοχές οι οποίες έχουν υψηλό επίπεδο ανεργίας, ψηλότερο από ό,τι στο μέσο όρο της Ένωσης. Βέβαια, η ιδέα αυτή μιας ε, σαφέστερης ε, παρέμβασης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ασφάλιση ενεργείας στην Ευρώπη κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που εκφράσαν και άλλοι ομιλητές. και για χώρες που μπορεί να ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα. Αλλά πάντως αν αναζητήσουμε έναν νέο τρόπο για του σταθεροποιητή. Θα πρέπει να κοιτάμε στις διαρθρωτικές πολιτικές, την απασχόληση, πολύ πιο, κατά τρόπο πολύ πιο προβεβλημένο από ό,τι μέχρι τώρα. Και με πρόσβαση στα κονδύλια και με προ... εμπροστοβαρή προσέγγιση. και με την δυνατότητα για προσωρινά μέτρα, όπως ε, μέτρα φορολογικού χαρακτήρα, παραδείγματι, ελάφρυνση στις περιοχές που υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Η δύσκολη στιγμή έχει φτάσει. Έχουμε πέντε λεπτά, μας δώσαν και ακόμα πέντε λεπτά οι διερμηνείς, αλλά έχουμε τις ερωτήσεις. Σέρκας, Εσάγια, Σορέντερ and Πώς εγώ βλέπω ότι είναι ένα εύκολο, ενδιαφέρον, απλό μοντέλο. Το θέμα της νομιμοποίησης του μοντέλου, ωστόσο, είναι κρίσιμο. Πώς νομιμοποιείς ένα ευρωπαϊκό, καθαρά ευρωπαϊκό μοντέλο, όπου αμοιβεοποιείται η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα σημαίνει ότι ο προπολογισμό της Ένωσης πρέπει να φτάσει στο 50%. Αυτό είναι απίθανο. Οι πολιτικές, οι πολιτικές προστασίας των νέων, εγώ 10 χρόνια μιλάω για μια ευρωπαϊκή επιδότηση νέων, τέλος πάντων κόντρα στο ρεύμα από ό,τι φαίνεται πηγαίνω, Υπάρχουν, μάλλον, τι πλονεκτήματα έχει ένα σύστημα που στηρίζεται σε ελάχιστο εισόδημα μάχης κατά της ανεργίας που δεν υποστηρίζεται και πολύ από την κοινή γνώμη σε σχέση με το με, με το μεταβιβάσεων και εξασφάλισης της ανεργίας. Mm-hmm. Κανείς δεν σκέφτηκε να εξετάσει στην Ευρώπη ένα πρόγραμμα κατά πολέμης ανεργίας αλλά που συνδέεται με ένα πολύ πιο αμφιλεγόμενο μοντέλο ως προς την δημόσια νομιμοποίηση. Η κυρία Σαΐα. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις είχα. Δεν έχουμε χρόνο. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν αφορά την αρμοδιότητα της Ένωσης στο θέμα αυτό. Στις σκανδιναβικές χώρες, Φερρυπίν, αυτά τα ταμεία τα χειρίζονται τα συνδικάτα. πώς θα μπορέσει να αλλάξει το σύστημα αυτό ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να αποκλείονται. Είχατε κάποιο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα αυτό. Τι λένε. Ο κύριος Φίσερ ανέφερε ότι τα εθνικά συστήματα είναι τόσο διαφορετικά τα επιδόματα σχετίζονται με το βαθμό, με, το μισθό. Και οι μισθοί είναι διαφορετικοί από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα που πρέπει να σκεφτούμε. Μια ακόμα ερώτηση. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ηθικού κινδύνου να πληρώνουν δηλαδή μέσω, τα εθνικά, μέσω των εθνικών ε, συνεισφορών τους οι εργαζόμενοι, ενώ η διαφορετική κατανομή να γίνεται από τα κράτη-μέλη. Αν ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα, γιατί να αλλάξουν τα εθνικά του συστήματα. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει ένας ε, ε, ελοχεύων κίνδυνος, η κυρία Σρέντορ. Το ότι διατυπώνω επικριτικές ή κριτικές ερωτήσεις σημαίνει ότι δεν μου αρέσει το σύστημα. Αντιθέτως, ασχολούμαι για καιρό μαζί του, γιατί δυόμιση χρόνια τώρα το κόμμα μας έχει εντατικά ε, ενσκύψει στο θέμα αυτό. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζει τους ανέργους και πώς ε, ένα σύστημα ασφαλιστικό στο οποίο δεν καταβάλει κανείς φορές μπορεί να ε, προσφέρει τα ασφάλιστρα, μπορεί να προσφέρει την, ε, τα, το, την, την ασφάλιση, μπορεί να λειτουργεί και πολλά άλλα ερωτήματα και επικριτικά τα οποία οδηγούν σε μια δυναμία να νομιμοποιήσουμε στα μάτια του κοινού ένα τέτοιο σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να πείτε εσείς πώς το βλέπετε στην πράξη. Μαρέ Σαχτιέ, Συμφωνώ και εγώ με τις ερωτήσεις των συναδέλφων και προσθέτω και μερικές επιπλέον. Πρώτον, έχετε μελετήσει το επίπεδο ανταπόκρισης ε, τέτοιων δράσεων για την καταπολέμηση ενεργεία σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, γιατί πάντα επανέρχεστε στο περιφερειακό επίπεδο και την έννοια της εγκύτητας. Δεύτερη ερώτηση, τι είδους ε, αναγνωσιμότητα για τον εργαζόμενο ή μάλλον τι είδους αιρεσιμότητα για τον εργαζόμενο και επίσης τι είδους ε, όρους συγκεκριμένα σκοπεύετε να ε, διατυπώσετε. Έχουμε πέντε λεπτά μόνο, άρα ο καθένας παρακαλώ να περιοριστεί σε ένα λεπτό την τοποθέτησή του για το θέμα της Ισπανίας Νομίζω ότι είναι σχετικά τα ερωτήματα. Λύσεις ουσιαστικές ε, δεν είναι αυτές, δεν είναι λύσεις λέει, για να βγούμε από την κρίση. Βοηθούν όμως ε, βραχυπρόθεσμα. Και αυτό σημαίνει να δοθούν βραχυπρόθεσμα λύσεις όταν όλο ο κόσμο κοιτάει την Ευρωζώνη, παραδείγματι, και περιμένει ένα ισχυρό μήνυμα που να δείχνει ότι πορευόμαστε μαζί. Αλλά επαναλαμβάνω δεν πρόκειται να λύσουν τα προβλήματα της κρίσης. Απλώς να απαλύνουν το, τον πόνο. Επομένως, ε, μεταφορές ε, από πλούσιες σε φτωχέ χώρες, όλα αλληλένδετα είναι και το βλέπουμε αυτό και στο γράφημα όπου η Ισπανία παρουσιαζόταν πάνω από το ε, μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να έχουμε ένα σύστημα για να έχουμε ένα μέσο όρο ανεργίας ως κριτήριο. Και έτσι θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιος είναι ο μέσος όρος. Πού θα βρισκόταν ε, η ανεργία της Ισπανίας αν δεν είχε τόσο βαθιά ύφεση. Θα ήταν χαμηλότερη ή πολύ χαμηλότερη. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να αντοπιστεί επακριβώς ε, το χρονικό πλαίσιο. Μπορούμε να πούμε ένα, μια πενταετία μέσα ανεργίας, σαν ορόσημο, σαν κριτήριο, και η χώρα θα συμβάλλει ανάλογα με αυτό το μέσο όρο της τελευταίας πεντέτειας. 12% πριν στην τελευταία πεντέτεια, η συμβολή. Ε, παραδείγματι, επί των μεικτών μισθών, δεν χρειάζεται να πούμε τα, ε, ΦΠΑ απαραίτητα ή κάτι τέτοιο, θα πούμε ότι ε, επί των ε, μεικτών μισθών αυτή θα οριστεί να είναι η συμβολή της χώρας. Και αυτό σημαίνει ότι αν παραμένει σταθερή ανεργία είναι μηδενική εισφορά της. Αν όμως αρχίζει διακυμάνεις άνω ή κάτω, τότε έχουμε την ανάγκη για ε, εισφορά και απόκληση η οποία θα διαρκεί όπως είπαμε πέντε χρόνια. Γιατί μετά τα πέντε χρόνια ο μέσος όρος πάλι μας προλαβαίνει. Έχει δηλαδή προσωρινό χαρακτήρα το μέτρο αυτό, δεν είναι σύστημα μεταφοράς κονδυλίων. Ένας άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σε πιο τοπικό επίπεδο και νομίζω πάλι ένα απλό σύστημα χρειάζεται. Δεν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο καταβάλλεται, θα μπορούσαμε να πούμε για τους πρώτους 12 μήνες ένα τμήμα το καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή όμως του συστήματος δεν έχει διαφορά για τον κοινωνικό εταίρο για αυτό το παράδειγμα της Γαλλίας τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Εφερειπίν στη Γαλλία γιατί την αντιπραγμάτευση του ΙΝΕΝΤΙΚ και του συστήματος αυτού κάλυψης με στο φθινόπωρο. τι της συζήτησης λοιπόν. αν δεν αφορά μια εναρμόνιση ή τι άλλο θα αφορά μια αντίληψη για το τι κάνουν τα άλλα κράτη. Αλλά και αυτό καλό το βρίσκω. Να συνεχίσω εκεί που σταματήσατε για το θέμα του κίνδυνου. Προφανώς υπάρχει κίνδυνος. Παντού, σε κάθε ασφάλεια περιλαμβάνεται κίνδυνος. Υπάρχουν πιθανότητες να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που να ενισχύει ή να μειώνει το κίνδυνο, αλλά υπάρχει ένα πιο βασικό θέμα. Είσαι, είμαστε στην, στο ΝΕ ναι μαζί. Μας ενδιαφέρει λοιπόν όλα τα μέλη της ΟΝΕ ναι να είναι αξιόπιστες οι διοικητικές ικανότητες. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει ήδη κάνει πολλά για να καλύψει θέματα διοικητικής ε, ικανότητας, ε, τμηματοποίησης της αγοράς, εργασίας. Ε, υπάρχουν θέματα που έχουν γίνει, θα γίνουν και άλλα. Μπορούμε να πούμε βέβαια ότι ένα ευρωπαϊκό σύστημα ανεργίας θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη συζήτηση αυτή. Να απαντήσω και στο ερώτημα του κύριου Σέρκας. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις του κυρίου Παράης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που σχετίζεται με αυτό μια πρόταση Σάδερλαντ και Άτκινς ενώ κοινωνικού οικονομολόγου για επιδόματα παιδιών που είναι, έχουν πολύ λιγότερο κυκλικό αντίκτυπο. Μπορεί να είναι προτάσεις κοινωνικής πολιτικής καλές, αλλά οι κυκλικές επιπτώσεις τους είναι μικρότερες. Δηλαδή η αντιμετώπιση της ανεργίας έχει μεγαλύτερα κυκλικά, κυκλικές επιπτώσεις. Μπορεί να συνεχίσουμε στα αγγλικά, μπορεί να μιλήσετε και σε άλλη γλώσσα. Να συνεχίσω αυτά που είπε ο κύριος Φίσερ, σύμφωνα με τον κύριο Σέρκας. Η ιδέα του ελάχιστου εγγυημένου μισθού είναι πρόταση κοινωνικής πολιτικής, όχι κυκλικής αντιμετώπισης. Το ελάχιστο πρόγραμμα εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή ή κακή ιδέα, αλλά είναι άλλο πράγμα. Για την ερώτηση της κυρίας Ισάια, συζητήσαμε με τα συνδικάτα στη Γερμανία, ενδιαφέρονται. Θα φανταζόμουν ωστόσο ότι δεν έχει ευρεία βάση εγώ θα έλεγα ότι τα πλεονεκτήματα στον χρόνο είναι για πάσα περίπτωση και υπάρχουν πλεονεκτήματα και για τους εργοδότες σε σχέση με τους, για τους εργοζόμενους σε σχέση με τους εργοδότες. Η αποδοχή ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να είναι υψηλότερη, γιατί σε όλες τις χώρες, τις χώρες της Νομισματικής Ένωσης έχει άτομα που κερδίζουν από το σύστημα, άρα θα γινόταν ελκυστικό και ευπρόσδεκτο για το κοινό. Σε αντίθεση με το δικό σας σύστημα που, αν καταλαβαίνω καλά, περιλαμβάνει ένα κεντρικό ταμείο που κατανέμει κονδύλια μεταξύ των μελών. Αυτό είναι άλλη ιδέα. Συμφωνώ μαζί σας ωστόσο ότι σχετίζονται, υπάρχει, υπάρχουν προβλήματα. Είχα ένα ολόκληρο slide που δεν είχα χρόνο να σας δείξω με τα προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε διαφορετικά συστήματα επιδοματών ανεργίας στην Ένωση. Άλλα σχετίζονται με τους καθαρούς μισθούς, ή περισσότεροι με τους ακαθάριστους μισθούς. Κάτι θα πρέπει να το ενοποιήσουμε από διεθνικά. Βεβαίω αυτό, όπω το είπε και ο κ. Φιλίππο, δεν είναι κάτι το βραχυπρόθεσμο, χρειάζεται χρόνο. και πολλά στοιχεία για να κρίνουμε τον αντίκτυπο της σταθεροποίηση και το πόσο, πόσα κονδύλια θα διανεμηθούν από χώρα σε χώρα. Με έναν προπολογισμό 50 δις ευρώ έχουμε κρίνει ότι μπορείς να εφαρμόσεις το παράδειγμα που είχα δείξει στη διαφάνειά μου με ένα χρόνο και 50% των προηγούμενων μισών. Αυτό είναι όμως μια πολύ έτσι γενικευμένη εκτίμηση. I fully acknowledge the, the problem. Αναγνωρίζω πλήρως ε, την ύπαρξη αυτών των προβλημάτων και γι' αυτό πρότεινα διάφορες εναλλακτικές λύσεις. και ε, δεν πρόκρινα μία παρέμβαση πλήρους κλίμακας ε, γιατί δεν είμαι σίγουρος θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά. Εγώ ήθελα να επικεντρωθούμε στις υπόλοιπες λύσεις. Αυτό το σύστημα συνεπάγεται μεταφορά πιστώσεων όχι ανάμεσα στις πλούσιες και στις φτωχές χώρες, αλλά ανάμεσα στις χώρες με χαμηλότερη ενεργεία και στις χώρες με υψηλότερη ενεργεία. Όταν ε, έλεγα ότι πρέπει να ισχύσει κάποια ερεσιμότητα, αυτό σχετίζεται και με τα κονδύλια. Δηλαδή, οι χώρες δικαιούχοι θα πρέπει να δεχτούν τους κανόνες ε, για τη χορήγηση των επιδομάτων που θα είναι κοινά συμπεφωνημένοι. Να μην δημιουργηθούν κίνητρα για τους ανθρώπους ώστε να παραμένουν άνεργοι γιατί αυτό συμβαίνει με τα επιδόματα ενεργείας. Εννοούσα πάντως, ε, και γι' αυτό σας μίλησα για αρεσιμότητα, ότι πρέπει αυτό να το προβλέψουμε στο πακέτο, στο σχεδιασμό του συστήματος. Άλλες δυνατότητες παρέμβασης. Ένα ταμείο της πολιτικής απασχόλησης θα μπορούσε να έχει καλύτερη χρηματοδότηση και πολύ χαμηλότερες μεταφορές ε, πιστώσεων και θα μπορούσε να δράσει πιο αποτελεσματικά σε περιφερειακό επίπεδο Οπότε δεν θα είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα της μεταφοράς των πιστώσεων. Θα ανέκυπταν κάποια τέτοια προβλήματα, όμως θα ήταν πολύ πιο light η εκδοχή και όχι τόσο απαιτητική για τον προϋπολογισμό και μεσοπρόθεσμα περιφέρειες που πλήττονται από την ανεργία θα υποφελούνταν περισσότερα. Σε περιοχές όπου είναι ευθύνουσα η οικονομική δραστηριότητα ή πολύ αυξημένη ανεργία των νέων, θα μπορούσαμε να γενικεύσουμε την εφαρμογή αυτής της αρχής και ε, στο μέλλον να τροφοδοτήσουμε το Ταμείο με υψηλότερα, ε, περισσότερα κονδύλια. Τρίτη εναλλακτική λύση, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Διοχετεύοντας για την περίοδο 2014-2020 περισσότερα κονδύλια στα διαρθρωτικά ταμεία και να αναδείξουμε σε βασικό κριτήριο το ποσοστό ανεργίας. Δηλαδή εκεί θα μιλήσουμε για τις διακοιμάνσεις σε σχέση με το μέσο όλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή άμα μια περιοχή υπερβαίνει ένα σχετικό ποσοστό ανεργίας πληρεί τα κριτήρια και άρα δεν χρειάζεται να συνεισφέρει τόσο πολύ αυτή η χώρα στον προϋπολογισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία. Φερρυπίν ή ε, θα εκταμιεύονται κάποια από τα κονδύλια και ξαναλέω ότι η ανεργία θα μπορούσε να είναι ένα κριτήριο για να χρησιμοποιούν με πιο ευέλικτο τρόπο ή με μπροστοβαρή τρόπο τα κονδύλια που τους αναλογούν τα κράτη-μέλη ή να ε, μειωθεί η συνεισφορά τους για τα διαρθρωτικά ταμεία. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό θα ήταν ένα καλό ε, σταθεροποιητή. Είναι εφικτή η εφαρμογή αυτή τη λύση και θα είχε άμεσο αντίκτυπο. Ένα ταμείο για την προώθηση των ενεργών πολιτικών ε, απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο είναι επίσης μια πολύ καλή ιδέα και πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα αυτή είναι μια λύση, να έχουμε το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά πρέπει να συζητηθεί ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ, Λύη Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ ε, πάρα πολύ και κυρίως τους διερμηνεί. Πρώτη φορά κάνω τόσο μεγάλη υπέρβαση. Δεύτερον, να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ. Ήταν συναρπαστική η αλλω σας ευχαριστω λυη προεδρος σας ευχαριστω ε παρα πολυ και κυριως του διερμηνεις πρωτη Είναι η πρώτη από μια μακρά σειρά τέτοιων ακροάσεων. Είναι πολύ καλό που εξετάζουμε διάφορες εναλλακτικέ λύσεις ε, και έχουμε και δύο πρωτοβουλίες. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα τεθεί ακριβώς αυτό το ζήτημα και θα βοηθήσουμε την Επιτροπή της δραστηριότητε που έχει σε αυτό το τομέα. Επίσης θα έχουμε μια υπηρεσία προσθέμενη αξία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εξετάζει τη δυνατότητα ανάληψη νομοθετική πρωτοβουλία για αυτό το ζήτημα ενδεχομένως κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο αλλά πάντως θα είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου στο μέλλον. Ξαναρχίζουμε στις 3.